Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Αν πάνε όλα καλά, και δεν υπάρχει και λόγος να μην πάνε όλα καλά, αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας στη διάρκεια αυτής της θητείας. Στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 3 θα πρέπει να προσθέσουμε και την έγκριση των πρακτικών της συνδυασής της 10 η και 13 η Φεβρουαρίου που είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες ε, στο φάκελό σας. Στο σημείο 4 η κυρία Ροτζούλη δεν θέλει να κάνει συζήτηση για συμβαστικές ε, τροπολογίες γιατί δεν κατάφερε να κάνει συμβαστικές τροπολογίες. Δεν μπορούμε ε, να ψηφίσουμε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα χωρίς συζήτηση, επομένως η κυρία Ροντζούλη δεν κατάφερε να κάνει συμβαστικές τροπολογίες. Θα περιμένουμε να έρθει για να ψηφίσουμε τις τροπολογίες χωρίς συμβαστικές τροπολογίες και θα γίνει συζήτηση επί του θέματος λίγο αργότερα. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως να είναι εδώ η συγγήτρια. Άρα το σημείο 4 θα συζητηθεί μετά το 5. Χωρίς τώρα περαιτέρω καθυστέρηση, σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 2 των εργασιών μας και έχω πέντε ανακοινώσεις να σας κάνω. Πρώτον, για πώληση. Δεν ξέρω αν έχουμε έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου εδώ. Δεν έχουμε. Το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί για την ανακοίνωση που θα σας κάνω εδώ σήμερα το πρωί. Μας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι αποφάσισε στο θέμα των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στο οποίο είχαμε μια ομάδα διαπραγμάτευσης, επικεφαλής ήμουν εγώ όπως συνήθως και ο εισηγητής είναι ο κύριος Δαρντά, ε, η το Συμβούλιο αποφάσισε να ε, εγκρίνει μονομερή δήλωση για το δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης έγραψα μια επιστολή στην Ελληνική Προεδρία, ε, διότι αυτή η δήλωση δεν είχε αναφερθεί σε καμία στιγμή των διαπραγματεύσεων. Ο πρέσβης μας απάντησε ότι η δήλωση περιλαμβάνει ε, τα όσα περιλάμβανε η δήλωση που είχαν κάνει τα κράτη-μέλη όταν ε, εγκρίθηκε η Γενική Προσέγγιση του Συμβουλίου. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για την ύπαρξη αυτής της δήλωσης και προκειμένου να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την πράξη αυτή πριν το τέλος της θητείας, η Πρόεδρος σας προτείνει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, αλλά να ζητήσουμε η δήλωση να μην δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα και το κείμενο να είναι όσο το δυνατόν πιο ε, κοντά στα όσα εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να συζητήσουμε βέβαια με την Ελληνική Προεδρία αυτή την κατάσταση, διότι όλοι όσοι γνωρίζουν πολύ καλά τα θέλατα συναπόφασης γνωρίζουν για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η δήλωση. Πολύ συχνά το Συμβούλιο προσπαθεί κατά αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει την ερμηνεία που θα μπορούσε να δοθεί στα κείμενα. εις βάρος των δικαιωμάτων του συνομοθέτη, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένως, θα πρέπει η δήλωση αυτή να ε, γίνει μόνο μετά από συμφωνία μεταξύ των δύο συνομοθετών. Και επειδή πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, συζητήθηκε ιδιαίτερα και στη θητεία μας ε, και στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου, το να υπάρχει αυτή η μονομερής δήλωση είναι απαράδεκτο. και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι ε, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ε, των κρατών μελών ε, θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο προαιρετικά ή υποχρεωτικά. Εμείς έχουμε πει ότι αυτή η συμμετοχή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Το Συμβούλιο έκανε μια ολόκληρη συζήτηση διότι ήθελε αυτή η συμμετοχή να είναι προαιρετική συζήτηση. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ήταν ένα κείμενο το οποίο ε, καταρχήν ικανοποιούσε τους πάντες ε, επειδή υπήρχε μια δημιουργική αφησιμία. Και εδώ το Συμβούλιο για άλλη μια φορά θέλει να επανέλθει για να επιβεβαιώσει κάτι το οποίο καταρχήν είχε δηλώσει με ικανοποίηση στο τριμερή διάλογο. Εμείς θεωρούμε ότι όλη αυτή η υπόθεση είναι απαράδεκτη και από την ε, γλώσσα του σώματός σας αντιλαμβάνομαι ότι έχω και την υποστήριξή σας για να συζητήσω περαιτέρω με την Ελληνική Προεδρία το θέμα αυτό για να το επιλύσουμε. Δεύτερη ανακοίνωση θα έχουμε μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή ε, Προπολογισμών για την ε, πρωτοβουλία απασχόληση για τους νέους. Προβλέπεται για την 1η Απριλίου από τις 10 έως τις 12.30 και όλοι οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής μας είναι προσκεκλημένοι φυσικά για να συμμετέχουν σε αυτή την ε, ακρόαση. Το πρόγραμμα θα σας αποσταλεί σε επόμενες ημέρες, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να σημειώσετε αυτή την ακρόαση Πρόκειται για μια πρωτοβουλία δική μα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει ισορροπία στην ακρόαση μεταξύ της Επιτροπής Προπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης να υπάρχει κατάλληλη εκπροσώπηση από πλευρά μα. Τρίτον, η πιο σημαντική σήμερα το πρωί ανακοίνωση στο τέλος της συνεδρίασης θα κάνουμε μια φωτογραφία με όλα τα μέλη της Επιτροπής και θα προσφέρουμε ένα ποτό έτσι για το τέλος της θητείας. Σημείο 4 για τη διερμηνία που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η σύνθεση της αντιπροσωπείας για τη Ρώμη τροποποιήθηκε μετά από κάτι αλλαγές που έγιναν την τελευταία στιγμή και επομένως θα υπάρχει αγγλική αντί της γερμανικής γλώσσας. Δεν ξέρω αν αυτό έχει συνέπειες στον προπολογισμό, αλλά είναι μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής και αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι κάποιο κόστος επιπλέον θα υπάρχει λόγω της αλλαγής ε, ε, που έκανε το ΕΛΚ. Πέμπτη ανακοίνωση. Ο φάκελος των θεμάτων της συνεδρίασης ε, διατίθεται πλέον μέσω της εφαρμογής e-meeting. Η Επιτροπή αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και νομίζω ότι στη διάρκεια αυτής της θητείας το Κοινοβούλιο ε, προχώρησε και έγινε μάλλον ηλεκτρονικό πλέον Κοινοβούλιο. Στο σημείο 3 πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά όλων αυτών των συνεδράσεων για τις οποίες δεν γνωρίζω για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν είχαμε εγκρίνει τα πρακτικά από τις 5 Δεκεμβρίου, 9 Δεκεμβρίου, 17 Δεκεμβρίου, 9 Ιανουαρίου, 22, 23 Ιανουαρίου, 3 Φεβρουαρίου, 12 και 13 Φεβρουαρίου. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Το σημείο 4 δεν έχετε ενστάσει για τα πρακτικά, επομένως εγκρίνονται. Το σημείο 4 είπαμε θα το κάνουμε μετά το σημείο 5. Πάμε στο σημείο 5. Δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την οδηγία 9671 για την απόσπαση των εργαζομένων και την εκτέλεσή της πιο συγκεκριμένα για τους ε, αποσπασμένους εργαζομένους στα πλαίσια παροχής υπηρεσίας. Να δώσουμε απευθεία το λόγο στην εισηγήτριά μας, την Ντανούτα Γιασλοβιέσκα. 27 Στις 27 Φεβρουαρίου δώσαμε τελική μορφή στις διαπραγματεύσεις ε, για την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Στις συνεδριάσεις μας, στις συναντήσεις μας είχαμε συζητήσει όλες τις πιο σημαντικές διατάξεις. 3, 9 και 12. Τρία χρόνια μετά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων κατέληξαν σε συμβιβασμό που φάνηκε, που είχε φανεί μάλλον, ε, αδύνατο να επιτευχθεί σε πολλές προεδρίες αλλά και σε πολλά ενδιαφερόμενα μέρη, stakeholder. Ως συνεισηγήτρια και συμπρόεδρος της διαπραγματευτικής ομάδος από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την υποστήριξη της έμπειρης συναδέλφου μας Προέδρου Περβάνς Μπερές. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους και, και όλες τις συναδέλφους μας, Στίβεν Χιούς, Νάντια Χίρς, την κυρία Σρέντερ, τον κύριο Χέντελ, Μίλαν Κάρμοφ, την κυρία Μακιντάια. Όλα λοιπόν αυτά τα πρόσωπα τα ευχαριστώ ιδιαίτερα καθώς και τις και τους συνεργάτες τους. Ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε είναι καρπός των προσπαθειών όλων μας. Και είμαι βεβαία ότι είστε όλοι οι περήφανε, όλες και όλοι οι υπερήφανες για το αποτέλεσμα. Από την αρχή, όταν αρχίσαμε δηλαδή την επεξεργασία της οδηγίας, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την νομική προστασία των εργαζομένων και ταυτόχρονα διαφάνεια για τους ε, εργοδότες που θα απαιτηθεί από αυτούς δηλαδή να εκπληρώσουν τις διατάξεις της οδηγίας για την προστασία των εργαζόμενων. Για να εκπληρούνται οι πιο βασικές ε, προϋποθέσεις, οι χώρες μέλη στην οδηγία υποχρεούνται να διαθέτουν μία επίσημη ιστοσελίδα με τις ε, διατάξεις και προϋποθέσεις για την απασχόληση καθώς και με τα περιεχόμενα των συλλογικών συμβάσεων και να δίνουν πρόσβαση σε οργανισμούς που θα δίνουν τις πληροφορίες για το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτή η ενιαία ιστοσελίδα θα είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών και για τους απασχολουμένους και για τους εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και για τους εργοδότες για τις υποχρεώσεις που ε, έχουν για να ε, εξασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι δε χώρες μέλη καλούνται να εποπτεύουν και να ασκούν έλεγχο. Η ε, διαδικασία κοινοποίησης πριν από την ε, απόσπαση. Η κοινοποίηση της απόσπασης του εργαζομένου με τις πληροφορίες σχετικά με την νομιμότητα της απόσπασης του συγκεκριμένου εργαζομένου στην χώρα υποδοχής και βέβαια με την κατάστασή του στην χώρα αποστολής. Τα δε μέτρα ελέγχου που έχουμε προβλέψει περιλαμβάνουν δράσεις που υποχρεώνουν τις εταιρείε να καθιστούν διαθέσιμα τα έγγραφά τους τα οποία εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απόσπασης και χρειάζονται και δύο συνομιλητές, contact persons, ένας που θα είναι, υποχρε... που θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση αλληλογραφίας και παροχή, και παροχή ε, ε, πληροφόρησης και ένα πρόσωπο ακόμη έξω από το εργοτάξιο για να εξασφαλίζει την επικοινωνία με τους ε, εκπροσώπους. Και πρέπει να περιγράφεται βέβαια και το είδος απασχόλησης για τον αποσπασμένο εργαζόμενο. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις παράνομης αυτοαπασχόλησης. για την εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων για την απόσπαση εργαζομένων. Και αυτό αποτελεί καταστρατήγηση του νόμου. Και στην ε, Ρώμη 1 προβλέπονται τα σχετικά μέτρα για την ένομη προστασία. Εάν λοιπόν πρόκειται για παράνομη περίπτωση απόσπασης, τότε είναι μία απόσπαση και θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ελεύθερη διακίνηση. Οι χώρες μέλη μπορούν να επεκτείνουν τον κατάλογο των μέτρων που προβλέπει η οδηγία έτσι ώστε να μπορούν να διώξουν αποτελεσματικά την παράνομη αυταπασχόληση μέσα στα πλαίσια της απόσπασης. Για να μπορέσει να αποφευθεί δε ο προστατευτισμός, οι χώρες μέλη καλούνται να προβλέπουν νέα μέτρα ελέγχου τα οποία θα είναι αναλογικά και αιτιολογημένα. Υποχρεούνται επίσης οι χώρε μέλη να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα νέα μέτρα ελέγχου τα οποία λαμβάνουν. Και βεβαίω να δημοσιεύουν τα μέτρα αυτά στην ενιαία εθνική ιστοσελίδα. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νέα μέτρα ελέγχου δεν σημαίνει ότι εγκρίνονται αυτομάτω η εφαρμογή τους. Οι χώρε μέλη θα πρέπει να έχουν ευθύνη στον τομέα της οικοδομής και να λαμβάνουν μέτρα για να αποφεύγεται, για να αποτρέπεται η παράνομη απασχόληση εργαζόμενων. Μπορούν να περιλάβουν και άλλους τομείς στην αλυσίδα υπερβολαβιών με την ευθύνη που βασίζεται στην αλληλεγγύη. Σε αλληλεγγύη ευθύνη δηλαδή. Οχτώ χώρες μέλη έχουν ήδη προβλέψει στη νομοθεσία τους την αλληλέγγυη ευθύνη. Και η οδηγία είναι έτσι γραμμένη ώστε να μην ανατρέπει το, το καθεστώς αυτό, το status quo αυτό. Οι χώρες μέλη συνεργάζονται για την δίωξη των παράνομων αποσπάσεων και είτε μέσω του κοινού συστήματος είτε διμερός πρέπει να μεταδίδουν τις σχετικές πληροφορίες για, για παράνομες αποσπάσεις. Ε, επίσης η οδηγία περιλαμβάνει, προβλέπει πρόστιμα στην περίπτωση παραβίασης του νόμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή και τη λειτουργία της οδηγίας και υπάρχει και ρήτρα επανεξέτασης που προβλέπει υποχρέωση της Κομισιόν να υποβάλει έκθεση μετά από μία τριετία. Ιδίω για τα στοιχεία που δικαιολογούν την απόσπαση, τα μέτρα ελέγχου, άρθρα 3 και 9, και την ελληνική ευθύνη του άρθρου 12, καθώς την, επίσης την αποτελεσματικότητα του συστήματος IMI για την επιβολή προστήμων. Και είναι επίσης απαραίτητο να, ε, εφόσον καταστεί απαραίτητο, να προταθούν ε, τροποποίησεις. Στη δική μου αξιολόγηση, όπως και στην αξιολόγηση των συναδέλφων μου, κατά την αξιολόγηση αυτή δηλαδή, το έγγραφο είναι ορθό, προβλέπει τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την ε, ένωμη προστασία των εργαζόμενων και για την διαφάνεια από πλευράς εργοδοτών, υποχρώνει τις χώρες μέλη να συνεργάζονται για την δίωξη των παράνομων αποσπάσεων. Εν τέλει θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκαρδίως και τους συναδέλφους μου και τους συνεργάτες τους, καθώς και τους συνεργάτες της Επιτροπής, καθώς και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και τις τέσσερις προεδρίες, Κυπριακή, Ιρλανδική, Ελληνική και Λιθανική, οι οποίες συνεργάστηκαν έτσι ώστε το έγγραφο να αποτελέσει την πηγή πραγματικά της πιο λογικής λύσης των προβλημάτων που θέτει η απόσπαση εργαζομένων. Σας συνιστώ και σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε τον συμβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Ευχαριστούμε για αυτή την ε, πραγματικά μεσατωμένη παρουσίαση του κειμένου. Ποιος θα ήθελε να παρέμβει? Τσιμινιούξ. Και Ρωσά Χιούς. Μετά Χάνταλ, Σχέντερ, Τσαπάουλη. Εντάξει, θα κλείσω ο ομιλητών. Παρακαλώ. Στίβεν Χιούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι είναι καλή συμφωνία. Θα ήθελα μάλλον να συμφωνήσω, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ. Θεωρώ ότι είναι κακή συμφωνία. Γιατί έχουμε ε, ρίξει πολλή δουλειά εδώ. Από αμέσω τη δεκαετία του 1990 παρακολουθούμε το θέμα. Ιδιαίτερα μετά την ε, δικαστική απόφαση λαβάλει το πριν από 7 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προσπάθειες που κατέβαλε και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας διαπραγμάτευσης, ε, στους χειώδεις συζητητές. Όμως θεωρώ ότι δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία, να συμφωνήσουμε επί ενός κειμένου που θα φέρει ε, ασφάλεια δικαίου ε, σε αυτό το ζήτημα. Πολλά κρίσιμα σημεία λοιπόν δεν έχουν διευθετηθεί κατάλληλα. Άμα δείτε στη συζήτηση που είχε γίνει μετά την Επιτροπή τη απασχόληση τον το προηγούμενο Ιούνιο και την ε, απόφαση που υιοθετήθηκε στο ΕΠΣΚΟ τα τέλη του χρόνου, αν τα συγκρίνετε αυτά με το κείμενο που συμφωνήθηκε στι 27 Φεβρουαρίου, θα δείτε ότι δεν υπήρξε κάτι ε, στη μέση όπω θα περίμενε κανεί από μια διαπραγματευτική διαδικασία. Το Συμβούλιο αρνήθηκε να διαπραγματευτεί επί των θεμελιωδών σημείων ε, ε, ε, του κειμένου. Υπήρχαν κάποιες βελτιώσεις στο άρθρο 3 και αλλού, όμως περισσότερο με προβληματίζει το άρθρο 9 και η έλλειψη προόδου στο άρθρο 12. Ανέφερα την έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο αναφέρεται ότι είναι καλή η συμφωνία γιατί στο άρθρο 9 για τα μέτρα ελέγχου είναι κλειστός ε, ο κατάλογος. Από την άλλη αναφέρεται ότι ε, είναι επιτυχία το ότι υπάρχει ανοιχτός κατάλογος. Δεν υπάρχει λοιπόν ασφάλεια δικαίου επ' αυτού. Είναι μια συνταγή ακριβώς για την αποτυχία, για την έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Και σίγουρα ε, θα, υπάρξει, θα αποτελέσει αντικείμενο νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το διάβασα πολλές φορές το κείμενο από τότε που το έλαβα. Νομίζω ότι το άρθρο 9 δίνει μια de facto ε, ένα κλειστό κατάλογο και θα δείτε ότι πολλά ε, σωματεία συμπεριλαμβανομένων των ε, ομοσπονδιών εργαζομένων συμπεριλαμβάνουν την απόσπαση και συμμερίζονται αυτή την άποψη. Στο άρθρο 12 δεν υπήρξε καμία μετακίνηση. Ένα κράτος μέλος μάλιστα εκβίαζε το Συμβούλιο, δεν ήθελε καμία μετακίνηση στο άρθρο 12, δεν υπήρξε καμία λοιπόν μετακίνηση στο άρθρο 12. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα είναι καλή η συμφωνία, δεν θα υπάρχει ε, ασφάλεια δικαίου που είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να επιτύχουμε. Κλείνοντα, Πρόεδρε, πρόκειται για προσωπική άποψη. Ναι, πράγματι παρακολούθησε τις διαπραγματεύσει, αλλά είναι προσωπική γνώμη αυτή που εκφράζω σήμερα το πρωί. Άλλα μέλη της ομάδας μου θα λάβουν διαφορετική θέση. Ευχαριστώ. Ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν το κεφάλαιο που είχαμε μπροστά μας, αλλά κάποτε ο Μπρέχτ είπε «Όδινεν όρος και έτε και μην». Ακριβώς αυτό ταιριάζει εδώ, στο αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας δύσκολη διαδικασία. Το αποτέλεσμα της ε, Επιτροπής ήταν αποδεκτό και μπορούσε κανείς να το χρησιμοποιήσει ως βάση για διαπραγμάτευση. Όμως, στον τριμερή διάλογο διαπιστώσαμε ότι από πλευρά Συμβουλίου βρισκόμασταν απέναντι στην ουσία σε ένα Συμβούλιο του Βατικανού. Δεν είχαν απολύτως καμία εντολή αυτοί οι τύποι να διαπραγματευτούν. Δύσκολο συμβιβασμός, ο οποίος κρατιόταν με παραμάνες, για να το πω έτσι δώσαμε, κάναμε μάλλον μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και δεν θα σας κρύψω, αναγνωρίζω ότι κάποιες βελτιώσεις μπόρεσαν να επιτευχθούν. Το σύνολο πάντως του αποτελέσματος δεν αποτελεί πραγματική βελτίωση και εξακολουθεί και είναι απαράδεκτο. Θα σας το εξηγήσω σε βάση πέντε παραδειγμάτων που θα συμφωνήσω σε ορισμένα και με τον Στίβεν Hughes και θα συμπληρώσω άρθρο 3, το οποίο άρθρο 3 δεν αποκλεί σε παράνομες αποσπάσεις τελικά να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας προέλευσης, δηλαδή ΡΟΜ 1. Και τελικά ένας να πληρώνεται χειρότερα από τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ασκήσαμε την κριτική εκεί. Είπαμε ότι η προηγούμενη κοινοποίηση δεν μπορεί να γίνεται στην περίπτωση αυτή, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν επίσης και αποτελεσματικοί έλεγχοι και με τον ανοιχτό κατάλογο είναι τόσο πολλοί περιορισμοί και τόσο ποικίλοι που στην ουσία ευνοούν προσπάθειες καταστρατήγησης του νόμου. Και το δόγμα της προστασίας του εργοδότη δεν ήθελε να το θίξει η ε, πλευρά του Συμβουλίου. Είναι λοιπόν κακή η ρύθμιση και μπαίνει και το ερώτημα πόσο θα, για πόσο θα εφαρμόζεται. Still stand, δηλαδή δεν θα προχωρήσει για μια πενταετία. Χρειάζεται τότε όμω την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να επανεξετάσουμε το θέμα και να επαναπραδιαπραγματευτούμε. Εγώ πάντω προτείνω και συνιστώ απόρριψη τη ρυθμίση που έχουμε μπροστά μα. Euh, Η κυρία Σρέντερ, μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Τσάμπα Όρη και άλλοι βουλευτές. Ελίζαμπεθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όποιος γνωρίζει το θέμα ε, γνωρίζει ότι νομικά είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση. Πάμε να ρυθμίσουμε εργασιακό δίκαιο σε ένα τομέα όπου στην πραγματικότητα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Ήδη από πλευρά συνθήκης είναι πολύ δύσκολο το θέμα. Και γι' αυτό είναι και δύσκολο και τόσο αμφισβητούμενο το γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να μειώσει, την, ε, να κάνει πιο ήπια την κατάσταση, αλλά έχασε. Εμείς μπορέσαμε να περάσουμε σημαντικά πράγματα ως Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε. Πρώτα, για το ερώτημα του ανοιχτού ή εξαντλητικού καταλόγου. Αν εξετάσετε το κείμενο, είναι σαφές ότι πρόκειται για ανοιχτό κατάλογο. Δηλαδή, οι χώρες μέλη, με άλλα λόγια, μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποια μέτρα θα λάβουν οφείλουν να τηρήσουν το πλαίσιο που θεσπίζει η συνθήκη, αλλά σε αντίθεση με την σημερινή κατάσταση, όπου το πλαίσιο το θεσπίζει στην ουσία με την ομολογία του το δικαστήριο, σε αντίθεση λοιπόν με αυτό, εμείς θεσπίζουμε τώρα το πλαίσιο. Είναι μία πρόοδος, δεν είναι τέλεια, αλλά δεν σημαίνει ότι πριν ήταν και καλύτερα. Οφείλω να το διαπιστώσω αυτό. Εγώ στην, ε, στο σημείο αυτό ήθελα να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο και κατέβαλα και μεγάλη προσπάθεια προσωπικά. Γνωρίζουμε πώς διεξήχθησαν οι τελευταίες ώρες των διαπραγματεύσεων, γνωρίζουμε και πού κόλλησε το θέμα και δεν μπόρεσε να προχωρήσει, πού εντοπιζόταν το πρόβλημα, πού και πώς στριμώχτηκε η Προεδρία στην γωνία, αν και καταρχήν ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει περισσότερα, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Και τι έχει συμβεί στα παρασκήνια. Αλλά εν ώψη του γεγονότος αυτού, εμείς παρόλα αυτά κατορθώσαμε να επιδείχνουμε κάποια μικρά βήματα προόδου και κυρίως ανατρέψαμε την προσπάθεια της Κομισιόν και αυτό είναι σημαντικό. Για το κεφάλαιο 3, εκεί είναι το θέμα η καταπολέμηση των εταιριών γραμματοκιβωτίου όπου μέχρι τώρα δεν υπήρχαν μέτρα για την καταπολέμησή τους. Δηλαδή, αν κάνουμε σύγκριση θα πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση ανάμεσα στο που ήμασταν ίσως αρχή τη θητείας μας. Δεν πετύχαμε βέβαια τα πάντα, αλλά στο άρθρο 3 νομίζω ότι πετύχαμε όντως τα πάντα. Σε ορισμένα πράγματα λοιπόν μπορέσαμε να περάσουμε αυτούς στις διατυπώσεις μας. Και ιδίω θέλω εκεί να θέσω και αυτό το λεγόμενο ερώτημα τι γίνεται με εκείνους που στην πραγματικότητα είναι αποσπασμένοι εργαζόμενοι, ψευδονίμως όμως. Εδώ η αιτιολογική σκέψη έχει δύο τμήματα και το δεύτερο τμήμα έχει τη μεγάλη σημασία και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι τέτοια ρύθμιση δεν έχει υπάρξει ποτέ ως τώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ρήτρα προστασίας δηλαδή για τα θύματα. Πρόκειται λοιπόν για πραγματική πρόοδο υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. Και οφείλω να το τονίσω αυτό, διότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει διάταξη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο που να περιλαμβάνει τέτοια διατύπωση. Αμέτρητες ώρες το συζητήσαμε το θέμα αυτό, αλλά εάν με ρωτήσει κάποιος πού ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των εργαζομένων, είναι εκεί ακριβώς. Στο σύνολό του το άρθρο 3 έχει πολλά σημεία όπου ενισχύονται τα μέτρα των εργαζομένων. Ω τώρα δεν υπάρχει καμία ρύθμιση μέσα στα πλαίσια τη ρύθμιση τη απόσπαση που να προβλέπει τόσο καθαρή ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Μιλούμε για ένα ντοσιέ που δεν βασίζεται στην ελευθερία διακίνησης, έτσι, αλλά στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Και γι' αυτό πρέπει και να δούμε ότι πράγματι εδώ βγαίνουν ενισχυμένοι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες και μάλιστα εκ του νόμου. Για δείξτε μου τον νόμο εκείνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου λέει ότι εδώ γίνονται πολλές καταχρήσεις. Στη δική μας νομοθετική πρόταση το γράφουμε σε τέσσερα σημεία. Ότι δηλαδή εδώ εντοπίζονται καταστρατηγήσεις του νόμου. Και γι' αυτό πρέπει να ρυθμίσουμε. Και αυτό οφείλουν να το κάνουν οι μέλη, διότι αυτέ έχουν τελικά την αρμοδιότητα. Πρόκειται για νόμους. Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα άλλο νόμο στην Ένωση που να τα λέει αυτά τα πράγματα τόσο καθαρά. Πάει να πει ότι εδώ πραγματικά θέσαμε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και να σκεφτούμε εάν πραγματικά όλα αυτά είμαστε διατεθειμένοι να τα πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων. Εν τέλει για το άρθρο 12, εκεί είχαμε μεγάλη δυσκολία. Προχωρήσαμε αρχικά πολύ φιλόδοξα και οφείλω να επενέσω εδώ τον Επίτροπο διότι έδειξε το θάρρος να ε, περιλάβει αυτή την ρήτρα περιευθύνης γνωρίζοντας ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να την κάνει δεσμευτική στο ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι έχουμε μόνο 8 χώρε μέλη που διαθέτουν στην νομοθεσία του τέτοια ρήτρα και μάλιστα και, ε, που βαίνει και μακρύτερα. Οι υπόλοιπε όχι. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε ρύθμιση κάπου όπου την αρμοδιότητα τη διαθέτουν οι χώρε μέλη και την αρμοδιότητα ελέγχου την διαθέτουν οι χώρε μέλη. Αυτό είναι γεγονό. Και ούτε θέλαμε καν να αλλάξουμε ε, το γεγονός αυτό. Διότι είχαμε τα 4 και 5 τη αρχική οδηγία. που περιγράφουν που εντοπίζονται οι αρμοδιότητε των ευμέρου κυβερνήσεων και τη Κομισιόν. Δεν θέλαμε να την αλλάξουμε. Με αυτή την βασική αρχή προχωρήσαμε. Ήταν λοιπόν εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία αφενό ε, να προωθούμε αυτού του φιλόδοξου στόχου και από την άλλη μεριά να γνωρίζουμε ότι οι χώρε μέλη δεν έχουν στο προστάσιό του ή ούτως ή άλλως τα μέτρα αυτά ελέγχου. Επιτύχαμε λοιπόν πολλά. Δεν αλλάξαμε ίσως απέναντι στο σχέδιο του Συμβουλίου, όμως διατηρήσαμε την πίεση. Επομένως και πριν από την ψηφοφορία μας εδώ στην Επιτροπή εξακολουθεί να, εφαρμόζεται, να εφαρμόζουμε πίεση στο Συμβούλιο για τη διαγραφή της 12. Είναι ένα πρώτο βήμα, μπορεί να προχωρήσει και επιτρέπει και ένα περιθώριο για εκείνες και εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν παραπέρα. Πολύ πιο εύκολα βέβαια θεσπίζεται η σχετική διάταξη αν έχουν ε, το σχετικό θεσμό στις νομοθεσίες τους και 28 χώρες μέλη. Όμως η κατάσταση όπου βρισκόμαστε σήμερα είναι τέτοια που 20 από τις 28 χώρες δεν διαθέτουν το θεσμό αυτό. Εφόσον γίνει αυτό λοιπόν, τότε θα είναι και πολύ πιο εύκολο να προχωρήσει, διότι έχουμε και ρήτρα επανεξέτασης, την οποία γράψαμε στην οδηγία. Το δικό μου συμπέρασμα εν τέλει είναι ότι υπό πάρα, πάρα πολύ δυσχερείς συνθήκες, υπό ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες, τα πολιτικά τα γνωρίζετε όλοι, δυσχέρειες που αντιμετωπίσαμε από όλες τις πολιτικές ομάδες διακομματικά, ωστόσο επιτύχαμε πολύ συγκεκριμένες νομοθετικές πρόοδους για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Αυτό είναι το συν. Πρόοδοι που έως τώρα δεν υπήρχαν στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Βέβαια δεν είναι τέλεια η οδηγία, ούτε και μπορεί να είναι τέλεια μέσα στα πλαίσια αυτής της κατάστασης μέσα από την οποία γεννήθηκε και κάτω από την πίεση και από τον τρόπο που διεξήχθησαν οι διαπραγματεύσεις και βεβαίως και τα όσα γίνονταν εκ παραλίλου με τις διαπραγματεύσεις Εφόσον λοιπόν τα συνυπολογίσω όλα αυτά, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι επιτύχαμε κάτι τι το οποίο αξίζει να το υποστηρίξουμε. Τώρα, εξ αντιθέτου, εάν το πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε σε ένα μελλοντικό κοινοβούλιο, όπου δεν θα έχουν αλλάξει οι συνθήκες πλαίσια, να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή το σχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης και βεβαίως και δεδομένων των δυσκολιών που προκύπτουν από το πλαίσιο των συνθηκών, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε στα επόμενα πέντε χρόνια να επιτύχουμε κάποια ουσιαστική πρόοδο απέναντι στο, στη ρύθμιση που έχουμε. Άρα, οι χώρες μέλη οφείλουν να δείξουν ότι είναι δυνατό να ασκηθούν οι έλεγχοι και αν κάπου φτάσουν σε κάποια όρια, τότε μπορούν μετά να τα προχωρήσουμε, γιατί θα έχουν την εμπειρία στο μεταξύ οι χώρες μέλη. Νομίζω ότι είναι μία οδηγία η οποία μπορεί να δεχθεί βελτιώσεις, μπορεί να δεχθεί παραπέρα επεξεργασία. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας καταρχήν κάποια εργαλεία και δεν είμαστε υποχρεωμένες να περιμένουμε την ομολογία του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ήρσος, συντονίστρια των φιλελεύθερων ε, ε, είναι κοντά μας. Θα ξανανοίξω λοιπόν το κατάλογο μιλητών για να τις δώσουμε το λόγο γιατί δεν έχει πάρει το λόγο φιλελεύθερος μέχρι τώρα. Τσαμαροή και μετά Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Αφενός θεωρώ ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες όλων όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το φάκελο, συμπεριλαμβανομένου ε, εισηγητή, συνεισηγητών και όλες τις ομάδες διαπραγμάτευσης που ε, τήρησε τα όσα είχε ήδη υιοθετήσει το Κοινοβούλιο η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, στηρίζει την ε, απόφαση, τη συμφωνία και, και νομίζω ότι αυτό θα εκφραστεί και κατά την ψηφοφορία. Εδώ αναφέρω την προσωπική μου γνώμη, δεν μιλώ ως ε, συντονιστής, εκεί αλλάζει η άποψή μου. Σημερίζομαι σε γραμμές τα όσα ανέφερε ο Στίβ προηγουμένως. δεν ε, πρόκειται για ρύθμιση, για διαθέτηση του τομέα. Είχαμε συζητήσει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή διατάξεων. Επιτύχαμε πρόοδο, σημειώσαμε πρόοδο σε αυτούς τους τομείς, όμως αυτό που θα θέλαμε, δηλαδή να έχουμε ξεκάθαρους, σαφέστατους και διαφανείς ε, κανόνες για την εφαρμογή, σε αυτό αποτύχαμε. Γιατί δεν έχουμε λιγότερους κανόνες, έχουμε περισσότερους. Πριν ε, καταλήξουμε σε αυτή την προκατακτική συμφωνία, λάβαμε σημαντικό αριθμό επιστολών από συνδικαλιστικές οργανώσεις, ε, οργανώσεις ε, εργοδοτών και ούτω καθεξής, που μας έλεγαν ότι αυτοί οι κανόνες δεν καθίστανται πιο σαφείς και ότι θα υπάρξει ε, νομική ασάφεια. Και όλες αυτές οι επιστολές μας οδήγησαν να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να καταστεί το κείμενο πιο σαφές και δεν κατανοούν γιατί πρέπει να δεχθούμε ε, το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση όταν υπάρχει τόση αβεβαιότητα. Ακούσαμε προηγουμένω ε, για το σημείο 9. Σύμφωνα με τον ε, Στίβεν, πρόκειται για εξαντλητικό κατάλογο, δεν είναι αρκετά ανοιχτό. Άλλοι, αντιθέτω, είπαν ότι πρόκειται για ανοιχτό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ε, διαμετρικά αντίθετες ε, απόψεις ε, για το ίδιο το σημείο. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι εντελώς αβέβαιη, γιατί λέμε ότι θα πρέπει αυτό να γίνεται με ανάλογο, αναλογικό και αιτιολογημένο τρόπο. Αλλά ποιος θα το κρίνει αυτό, θα είναι το δικαστήριο, θα κάνουμε μακροσκελέστατες συζητήσεις και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα. Δεν υπάρχει έλεγχος, πραγματικός έλεγχος. Οποιοςδήποτε, οποιαδήποτε αρχή μπορεί να πάρει μέτρα χωρίς κανέναν έλεγχο. Πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τους προβληματισμούς όσων είναι υπέρ ε, της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Άλλοι ανησυχούν για την εσωτερική αγορά, λένε ότι θα υπάρχουν πιέσεις στην εσωτερική αγορά και ότι θα είναι πολύ δύσκολο να ε, επανορθώσουμε την κατάσταση. Θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρή αβεβαιότητα σε νομικό επίπεδο και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να αφήσουμε ανοιχτό αυτό το διάλογο, να μην κλείσει αυτό το ζήτημα σε πρώτη ανάγνωση αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει δεύτερη ανάγνωση. Ορισμένοι λένε ότι οι ευρωσκεπτικιστές ε, θα είναι πιο ισχυροί στην επόμενη θητεία και δεν θα είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μας ε, για να βρούμε, να καταλήξουμε σε καλές συμφωνίες. Όχι, εγώ δεν ανησυχώ. Όπως και να έχει, πρέπει να προσδιορίσουμε ότι ακόμα και αν υπήρξε πρόοδος, ε, αν κάναμε θετικά βήματα, έχουμε βρει καλύτερους ορισμούς, σε ό,τι αφορά την παράνομη αυταπασχόληση και καταφέραμε να το δεχτεί το Συμβούλιο. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι πετύχαμε σε ό,τι αφορά ε, το να έχουμε έναν ε, καλύτερο προσανατολισμό για το ποιος ε, πρέπει να κάνει τι, ποια θα είναι τα νομικά μέσα που θα έχουμε. Σε αυτά λοιπόν τα σημεία δεν καταφέραμε να βρούμε μια κατάλληλη λύση. Δεν έχουμε πετύχει λοιπόν τους βασικούς μας στόχους, όπως και να έχει όμως σημειώθηκε πρόοδος και αυτό είναι θετικό. Ελπίζουμε να βρούμε ακόμα καλύτερες λύσεις στη συνέχεια σε ό,τι αφορά ε, τα σημεία από τα οποία υπάρχει διαφωνία και υπάρχει αντίφαση μεταξύ των θέσεων ε, των εργοδοτών και των εργαζομένων. Υπογραμμίζω ότι υπάρχει διχογνωμία απόψεων, ακόμα και στο ιστορικό του ΕΛΚ. Η πλειοψηφία των συναδέλφων μου θεωρούν ότι είναι αποδεκτή η συμφωνία και θα ψηφίσουν αναλόγως. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αλεχάνδρο Θέρκας και μετά η Νάντια Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, οι σοσιαλιστές παρακολούθησαν το θέμα αυτό με ανησυχία η οποία είναι ιστορικής φύσεως, όπως είπε και ο εισηγητής ο Στίβεν Χιούς, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για το έργο του, για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν για ένα θέμα το οποίο για μας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και εξακολουθεί να μην μας ικανοποιεί σχεδόν καθόλου. Μας ανησυχεί διότι αφορά την απόσπαση εργαζομένων ε, για ε, σκοπούς παροχής υπηρεσιών. Το θέμα αυτό, το οποίο αναφέρθηκε και ε, λόγω της οδηγίας Bolkenstein, τότε όταν μας απασχόλησε η βασική ανησυχία του Κοινοβουλίου ήταν να εγγυηθούμε όχι μόνο στου εργαζόμενου, αλλά και στι επιχειρήσει ότι δεν θα υπάρχει σε καμία περίπτωση κοινωνικό dumping με πρόσχημα την απόσπαση εργαζομένων. Οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι όταν θα βρίσκονταν σε μια άλλη χώρα μέλο, θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα ε, της χώρας ε, ε στην οποία θα έχναν κανένα κοινωνικό και εργασιακό δικαίωμα. Όταν συζητήθηκε η οδηγία Bolkenstein, έγινε σαφές ότι η απουσία κοινωνικού dumping θα μπορούσε να εγγυηθεί να, ε, ε, για τους εργαζομένους και να μην υπάρχουν ε, απάτες σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα μπορούσε να γίνει μέσω της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άλλαξε τη νομική αξία των συμβάσεων και άλλαξε τελείως ε, τα εργασιακά δικαιώματα και καθόρισε ότι οι οικονομικές ελευθερίες είναι υπεράνω των εργασιακών δικαιωμάτων. Και έπρεπε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι είναι τεράστια η κοινωνική ανησυχία. Υπάρχουν χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, στις οποίες ε, χιλιάδες εργαζόμενοι με το πρόσχημα της απόσπασης παρέχουν υπηρεσίες δύο ή τρεις φορές ε, με μισθου συγγνωμη συγγνώμη, δύο-τρει φορέ λιγότερου από ό,τι γίνεται. Και υπάρχουν ε, επιχειρήσει ε, φάντασμα που εδρεύουν σε φορολογικού παραδείσους, στο οποίο δεν υπάρχει καμία ρύθμιση και υπάρχει πλήρες νομικό κενό. Εκατοντάδε χιλιάδε λοιπόν εργαζόμενοι από φτωχότερε χώρε ή από χώρε ε, λιγότερο ανεπτυγμένε παρέχουν υπηρεσίε σε συνθήκε, οι οποίε είναι άδικες και ορισμένες φορές ομοιάζουν και σε συνθήκε σκλαβιά. Και στι χώρε τι οποίε η την νομοθεσία, ε, δίνεται η αίσθηση ότι ε, γίνεται εις βάρος τους όλη αυτή η διαδικασία. Πρόκειται λοιπόν για πολύ άδικες συνθήκες και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους. Το πρόβλημα όμως είναι η Οδηγία 96 και μάλιστα οι συνθήκες οι οποίες δεν έχουν καθορίσει σαφής, ε, σαφέστατα την ισορροπία μεταξύ ελευθεριών και δικαιωμάτων. Η οδηγία λοιπόν την οποία συζητούμε, δυστυχώς ε, δεν είναι ικανοποιητική για την ομάδα, διότι μια διοικητική οδηγία που αφορά τις ε, δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί να θέσει ε, επί ίσης ώρες τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που θέλουμε. Όταν ο κύριος ε, Μπαρόζο ε, ανέλαβε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του θέσαμε ως προϋπόθεση να συζητηθεί η οδηγία 9671. Δεν τήρησε τα όσα του είπαμε και μας έδωσε απλώς αυτή τη διοικητική οδηγία. Είναι με ένα βήμα προς τα μπρος, διότι σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία ε, δημιουργεί η κακή αρχιτεκτονική δομή της οδηγίας υπάρχουν και τα ε, προβλήματα ε, τα οποία δημιουργούν οι εικονικές εταιρείες οι οποίες ανέσχυντα δημιουργούν προβλήματα. Το είπε και η πρόεδρος, ε, η συνάδελφε και η συγγήτρια, προσπαθώντας ε, να σταματήσουν την απάτη, ε, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Και οι σοσιαλιστές θα ήθελαν να δηλώσουν σήμερα ότι για μας αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ολοκληρώνεται σήμερα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχει καν τεθεί διότι δεν έχει τεθεί προς συζήτηση η βασική οδηγία, η ερμηνεία των συνθήκων που οδηγούν ασυμμετρίες μεταξύ ελευθεριών και δικαιωμάτων. Και η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι αυτό κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Δημιουργεί πολιτικά προβλήματα πάρα πολύ μεγάλων διαστάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός, αυξάνεται η ξενοφοβία, αυξάνεται ο ρατσισμός και το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα ήθελα λοιπόν να είναι σαφές ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ομόφωνα οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές ε, αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να αλλάξει αυτή η οδηγία και να αλλάξει η ασυμμετρία που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Κατόπιν έρχεται το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα και θα ψηφίσουμε. Πρόκειται για μια σαφώς διοικητική οδηγία και ισχύει για, 18, για 28 χώρες που έχουν τελείω διαφορετικά δικαιώματα και τελείω διαφορετική νομοθεσία. Ακούσαμε την άποψη των συναδέλφων που θεωρούν ότι στις χώρες τους η οδηγία αυτή βελτιώνει ακόμα και, και λίγο, αλλά έστω και λίγο δημιουργεί κάποια βελτίωση. Επομένως θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε μια θετική ψήφο. Υπάρχουν συνάδελφοι στην ομάδα μου που θεωρούν ότι η οδηγία αυτή είναι αδιάφορη, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, διότι δεν θα αλλάξει η πραγματικότητα στη χώρα τους. Και υπάρχουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι ακολουθώντας υποδείξεις και κριτήρια των εθνικών συνδικάτων, θεωρούν ότι αυτή η οδηγία θα αποτελέσει ανάχωμα στην απάντηση στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Επομένως, ε, οι σοσιαλιστές θα ψηφίσουν με τρεις τρόπους. Θα υπάρχει ομοφωνία στην ουσία του θέματος, αλλά ε, η οδηγία δεν πάβει να είναι μια σαφώς διοικητική οδηγία που δεν δίνει κανένα επιπλέον δικαίωμα και απλώς καθορίζει κάποιους ελάχιστους κανόνες για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν κανένα τρόπο ελέγχου και επομένως ε, αυτά όλα θα τύχουν τη θετικής μας ψήφου. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θεωρώ ότι καλά θα κάνει το Κοινοβούλιο να τίνει ευήκο νου στα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Και αυτό θα το δούμε στις 25 Μαΐου. Θα δούμε πώς θα αυξηθεί η αίσθηση κατά της Ευρώπης και ε, πώς ε, χιλιάδες εργαζόμενοι θα νιώθουν ότι δεν τους εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, για τους οποίους έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να επιτρέπουν απόλυτη ελευθερία στην αγορά, Ολισμονώντας ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Εγώ προσωπικώ θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητική κατάσταση, καθόλου ικανοποιητική και σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη οδηγία δεν θα επιλύσει το πρόβλημα. Οι σοσιαλιστέ θα ψηφίσουν κατά συνείδηση και επομένω ε, θα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει ο καθένα ελεύθερα στην ομάδα μα. Ευχαριστώ. Έχω κλείσει το κατάλογο ομιλητών. Μόνο οι σχοιώδει και οι συντονιστέ ε, έχουν μπει. Η Νάντια Χίρσο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα να ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας των φιλελευθέρων την εισηγήτρια για την ε, πολύ θετική και επικοδομητική συνεργασία ημέρες αμέτρητες καθίσαμε και εργαστήκαμε και είδαμε καθαρά ότι δεν είναι απλό το θέμα, όμως όλοι κατέβαλαν, όλες και όλοι κατέβαλαν προσπάθειες για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και είμαι πεπισμένη ότι τώρα έχουμε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα πλέον όπου ε, όλοι μας νομίζω μπορούμε να το αποδεχτούμε. Υπήρξαν βελτιώσεις. Η αφετηρία από την οποία ξεκινήσαμε ήταν τέτοια που διαπιστώσαμε ασφαλώς ελλείψεις, διαπιστώσαμε προβλήματα, διαπιστώσαμε καταστάσεις λόγω της ε, υφιστάμενης ρυθμίσεως που ήταν απαραίτητο να καλυφθούν. Εάν κάποιος θέλει να βελτιωθεί η κατάσταση, έστω και με μικρά βήματα, υπάρχουν όμως βελτιώσεις τότε, εφόσον το θέλετε αυτό, πρέπει να υποστηρίξετε την έκθεση και την έκβαση των τριμερών διαλόγων. Διότι ασφαλώς υπάρχει ένα συν υπέρ των εργαζομένων, αλλά υπάρχει και περισσότερη διαφάνεια για τις επιχειρήσεις. Και αυτά είναι δύο σημαντικά θέματα, δύο σημαντικά στοιχεία. Αν περιμένουμε μέχρι ότου γίνουν όλα τέλεια, εμείς ως Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα φτάναμε, αν περιμέναμε πάντα το τέλειο, ποτέ εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ και ειδικά η αγορά εργασίας στην Ευρώπη είναι τόσο πολύ σε κίνηση που νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να πούμε με ήσυχη συνείδηση ότι επιτύχαμε πραγματικά μια βελτίωση υπέρ των εργαζομένων αλλά και των επιχειρήσεων. Υπάρχουν βελτιώσεις, υπάρχουν και οι δυνατότητες να εισαχθούν έλεγχοι από πλευράς χωρών μελών, να ανακοπεί το dumping των μισθών χωρίς ταυτόχρονα να ξεφύγει από τα όρια η γραφειοκρατία θεωρώ ότι οι χώρες μέλη είναι πολύ διαφορετικές και το έχουμε λάβει υπόψη αυτό, ώστε μπορώ να πω εξ ονόματος της φιλελεύθερης ομάδας ότι το αποτέλεσμα δεν είναι τέλειο, αλλά ωστόσο έχει επιφέρει βελτιώσεις. Και όποιος επιθυμεί σήμερα να επιφέρει βελτιώσεις, ιδίως υπέρ των εργαζομένων, που πράγματι είναι ο πιο ασθενής κρίκος συνήθως μέσα στην αλυσίδα της εργασίας, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπερψηφίσει το κείμενο. Και εμείς ως φιλελεύθεροι και φιλελεύθερες αυτό θα πράξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, φτάνουμε στο τέλος του καταλόγου μελετών. Ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, αλλά και της ομάδας διαπραγμάτευσης, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και το σύνολο των σκιωδών εισηγητών που είχαν δύσκολο έργο, υπό δύσκολες συνθήκες εργάστηκαν. Είδαμε ε, πώς ε, έτυχε επεξεργασία ε, η, η εντολή συγγνώμη, αυτής της ομάδας. Θα ήθελα μόνο να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, το είπα και στην ομάδα διαπραγμάτευσης, το λέω και εδώ δημοσίως, στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, ότι σε αυτό το φάκελο, όπως και σε άλλους, είδαμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο όταν ε, οι όροι συμφωνίας με το Συμβούλιο τυχαίνουν διαπραγμάτευση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Μπορεί να υπάρχει μια γενική προσέγγιση που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, που δεν ισχύει και πάντα, όμως ε, όταν ε, έχει καθοριστεί αυτή η γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο, το περιθώριο ευελιξία ε, στο Συμβούλιο για να επιτρέψει ε, μια προσέγγιση με το Κοινοβούλιο, όταν δεν ε, ταυτίζονται οι θέσεις Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, εκεί υπάρχουν λοιπόν δυσκολίε. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο το σύνολο της ομάδας διαπραγμάτευσης, με πραγματικά την συμβολή κάθε μέλους της ομάδας, επέτρεψε την βελτίωση του κειμένου του Συμβουλίου. Υπήρξαν νέες ε, διατυπώσεις που εισήχθησαν και σημεία προβληματισμού που εξομαλύνθηκαν μέσω των διαπραγματεύσεων επί της ουσίας και επί της διατύπωσης. Το τρίτο στοιχείο που θα ήθελα να θίξω είναι ότι στη διαδικασία της συναπόφασης η ισορροπία μεταξύ των εταίρων είναι σημαντικό στοιχείο. Και βλέπουμε ότι εδώ βλέπουμε την αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου, την ε, σαφήνεια της εντολής μας και η πυγμή με την οποία διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις ήταν σημαντικό στοιχείο. Επί της ουσίας έχουμε πει πολλά στοιχεία σήμερα. Είπαν κάποιοι στην αρχή της εντολής, μετά ε, τις αποφάσεις Λαβά και Λίκινγκ, για το διακύβευμα της αναθεώρησης της οδηγίας ή σε ό,τι αφορά την ισορροπία που έχει επιτευχθεί με τις ε, ε, συνθήκες, θεωρώ ότι όλα αυτά μένουν ανοιχτά για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ισορροπία τη συνθήκη. Αυτό παραμένει ανοιχτό ζήτημα. Εφόσον ε, δεν μπορούμε να έχουμε βεβαίως διπλή νομική βάση για ε, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και όταν θα έχουμε μια τέτοια πρωτοβουλία μια, ε, βλέπουμε την ανισορροπία που υπάρχει στο νομικό πλαίσιο όπως αυτό έχει οριστεί. όπως και η πλειοψηφία, ελπίζω και η Επιτροπή να συμφωνήσει και όπως ε, συνεπέρανε και ε, η ομάδα διαπραγμάτευσης, ε, σημειώνεται πρόοδος, σημαντική πρόοδος, σε έναν δύσκολο φάκελο που μας απασχόλησε καθ' όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την εξέταση αυτού του σημείου της μέσας διάταξης. Θα ψηφίσουμε σε λίγο για τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου. Αλλά όπως ανέφερα και στην έναρξη των εργασιών μας, ε, θα περάσουμε τώρα στο σημείο 4. Θα γίνει η συζήτηση για την έκθεση που αφορά την πρόταση οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 2008-94 και 2009-38, 2002-14, 98-59 και 2001-23. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρονσούλη Επί της αρχής, ε, με αυτό το σημείο θα μπορέσουμε να ενημερωθούμε για τις ε, συμφωνίες ε, τις συμβιβαστικές. Δεν υπάρχουν συμβαστικές τροπολογίες, επομένως έχουμε αυτή την μοναδική ευκαιρία όπου δεν υπάρχει μοναδική περίπτωση, μάλλον μοναδικό φαινόμενο, όπου καμία συμβιβαστική τροπολογία δεν υποβάλλεται στα μέλη της Επιτροπής. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Ρονσούλη. Ωραία. Βλέπω ότι αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια ο τρόπος με τον οποίο ε, διαχειρίζεστε την Επιτροπή, ε, κυρία Πρόεδρε, άλλαξε, διότι δίνετε και ψευδείς πληροφορίες. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν θέλησαν να υποβάλω συμβαστικές τροπολογίες. Ήθελα σίγουρα να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων μου. Αλλά ο συμβιβασμός, αλήτη συμβιβασμός, διότι πρέπει κάποιοι να προσπαθήσουν να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση ή να βρουν κάποια κοινά σημεία ώστε να υπάρξει μια κοινή κατεύθυνση. Ίσως όχι όλοι μαζί, ίσως όχι απόλυτη ταύτιση, α, καλείται όμως συμβιβασμός διότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, εκατέρωθεν ε, διαθέσεις να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξε κανένα κοινό σημείο και οι τροπολογίες που πρότειναν οι άλλες πολιτικές ομάδες πήγαιναν σε εντελώ αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με το όσα έκανα εγώ σε αυτή την έκθεση. Αυτή είναι η εξήγηση και όχι το γεγονός ότι δεν θέλησα να σεβαστώ τους συναδέλφους μου ή δεν ε, σεβάστηκα το έργο των υπολείπων. Και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό διότι δεν μ' αρέσει να περνάει κάτι τέτοιο ως μήνυμα. Πάντα σεβάστηκα το έργο των υπολείπων, ακόμα και αν είχαν αντίθετη άποψη ή αντίθετες ιδέες από μένα. Εδώ όμως, επειδή πρόκειται για μια έκθεση η οποία κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τους εργοζομένους και όσον αφορά δηλαδή τις θέσεις εργασίας, αλλά και για όσους δημιουργούν θέσεις εργασία, είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχουν σημεία ταύτιση, δεν μπορούμε να έχουμε συμβιβασμούς. Αυτό εν είδη εξήγηση σε σχέση με τα όσα μόλις είπατε και τα οποία στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνονται καθόλου στα όσα συνέβησαν. Έχω κάνει αρκετές παρουσιάσεις για το θέμα αυτό. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω άλλο την ψηφοφορία για να είμαι ειλικρινής. Να επαναλάβω και πάλι ότι η ναυτική δεν έχουν ακόμα ε, την ε, ε, ασφάλεια που τους πρέπει. Αυτή η δήλωση είναι απόλυτα λανθασμένη όμως. Υπάρχουν στα 28 κράτη-μέλη δεσμεύσεις οι οποίες διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων του τομέα και ορισμένες φορές οι κανόνες αυτοί εγγυούνται πολύ καλύτερα και με πολύ πιο σύγχρονο τρόπο τα όσα προβλέπουν οι πέντε οδηγίες. Γι' αυτό ακριβώ και δεν συμφωνούσαν να συμπεριληφθούν και οι ναυτικοί στον τομέα αυτό στις οδηγίες θα μπορούσαμε ίσως εδώ στη διάρκεια τη ηττίας να προσπαθήσουμε να έχουμε οδηγίε οι οποίες να εγγυώνται περισσότερα πράγματα και να προσφέρουν περισσότερα στους ναυτικούς. Αλλά θεωρώ ότι είναι δημαγωγία και ε, κοντόφθαλμο να θεωρούμε σε αυτή την τόσο σημαντική ιστορική στιγμή, απλώς και μόνο για προεκλογικούς σκοπούς, να αποφασίσουν να μην ακολουθήσουν την πιο αντικειμενική γραμμή που είναι υπέρ και των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών. Πραγματικά ε, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικά αυτά που προτείνω. Οι τροπολογίες ε, προφανώς έχουν συνεισφέρει στη βελτίωση του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διασφαλίζοντας και στους ναυτικούς την καλύτερη κοινωνική ασφάλιση και εγγυόμενη και το... Ε, δικαίωμα σε κατάλληλη προστασία και επίσης ε, και κατάλληλη ανταγωνιστικότητα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα ε, αυτού του ε, θέματος. Θα χαθεί η ανταγωνιστικότητα των εργοδοτών ε, υπέρ ε, σκαφών που χρησιμοποιούν σημαίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όλες οι θέσεις οι εργασίας οι οποίες δημιουργούνται χρησιμοποιώντας καινοτόμα στοιχεία και μειώνοντας τη γραφειοκρατία γίνεται ε, υπ' αυτούς του όρους. Εάν ένας εφοπλιστής βλέπει να του επιβάλλονται κανόνες που δεν το προστατεύουν σε διεθνές επίπεδο και δεν διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και αυτό σημαίνει ότι το, ως άμεσο αποτέλεσμα θα έχουμε πάυση των εργασιών τους, σημαίνει ότι χάνονται θέσεις εργασίας και επομένω δεν προστατεύουμε τους εργαζομένους. Σε περίπτωση που γίνεται μεταφορά της επιχείρησης, πώληση, ο ναυτικός έχει δικαίωμα να αποφασίσει αν θέλει να πάει στη μία χώρα ή στην άλλη, δεν υποχρεούται και να πάει στο νέο, στη νέα επιχείρηση και πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους. Δεν θα ήθελα να προτείνουμε πράγματα τα οποία δεν γίνεται να πραγματοποιηθούν. Θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους, να μην υποκύπτουμε σε προτάσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και προεκλογικές υποσχέσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα προστατεύσουν περισσότερο τους ναυτικούς που ούτως ή άλλως προστατεύονται. Συγγνώμη για την παθιασμένη ε, παρουσίασή μου, αλλά έχω κάνει πολλή δουλειά και πραγματικά θα με δυσαρεστούσε ιδιαίτερα να πάει χαμένο όλο αυτό το έργο. Κυρία Εισηγήτρια, ε, διαφωνώ απολύτως με την ερμηνεία που δώσατε στα λόγια μου. Ανέφερα ότι δεν υπήρξε συμβαστική τροπολογία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού, πού είναι οι συμβαστικές τροπολογίες, δεν υπάρχουν. Δεν μπορείτε λοιπόν ε, να διαφωνήσετε μαζί μου από αυτού. Το λόγο έχει η κυρία Μπαλτοτσίνο. Ποιο άλλος θέλει να πάρει το λόγο μετά την κυρία Μπαλτοτσίνο. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά εκπλήσω με ιδιαίτερο μετά όσα είπε η συγγήτρια, κυρία Πρόεδρε, γιατί ούτε καν συναντηθήκαμε. Ούτε καν είχαμε χρόνο. Δεν είχε χρόνο η συγγήτρια να γίνει τουλάχιστον μια συζήτηση πόσο μάλλον ε, να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Ναι, βεβαίως. Ιστορική στιγμή για όλους λέτε. Λέτε ότι είναι ιστορική στιγμή για όλους. Ναι, είναι. Για ποιον όμως είναι. Γιατί τώρα είναι στιγμή και πραγματικά πιστεύουμε σε μια κοινωνική Ευρώπη και πρέπει να προστατεύσουμε και τους ναυτικούς. Δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε από την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ναι, ναι, έτσι είναι. Και αφήστε με να ολοκληρώσω γιατί εγώ δεν σας διάκοψα. It is not true that our compromise that our uh, proposal... Δεν είναι αλήθεια ότι οι συμβαστικές προτάσεις ε, είναι επιζήμιες για την ανταγωνιστικότητα. Για παράδειγμα, κυρία Πρόεδρε, Μακάρι να είχαμε καταφέρει να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση για να συμπεριληφθούν και τα δικαιώματα των ναυτικών στι υφιστάμενε οδηγίε. Έτσι θα υπήρχε η μεταχείριση, λαμβάνοντα υπόψη και τι ειδικέ συνθήκε που ισχύουν για τι επιχειρήσει του κλάδου. Αλλά ε, ούτε καν συζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε σήμερα, γιατί δεν επιβλήθησαν οι συμβαστικές τροπολογίε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικαιροποιηθούν αυτέ οι οδηγίε και να αναρωτηθούμε πώ μπορούμε να δικαιολογήσουμε ακόμα το γεγονό ότι αποκλείται αποκλείονται οι ναυτικοί από αυτές τι οδηγίες. Ακόμα και αν ακολουθήσουμε μια πολυλογική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα και λαμβάνοντας υπόψη νόμους και συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους, το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ε, την ε, ε, Σύμβαση για τη Θάλασσα και ταυτόχρονα να σεβαστούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και να επιμένουμε οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν σε αποφάσεις όσον αφορά φερεγγιότητα επιχειρήσεων, πώληση σκαφών δεν έγινε καμία προσπάθεια για συμβιβαστικές προτάσεις από την εισηγήτρια. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε καρποφόρες συζητήσει. Στην πραγματικότητα δεν είχαμε καν συζητήσει. Η εισηγήτρια ακολούθησε μια πολύ πιο ακραία θέση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να παραμείνουν οι εξαιρέσει, αγνοώντας ε, σχεδόν αποκλειστικά ε, τις εξελίξεις μεταξύ των κοινών εταίρων και την ύπαρξη ε, σύγχρονων μορφών επικοινωνία που επιτρέπει στους ναυτικούς να συμμετέχουν και σε και να συμμετέχουν σε συμφωνίες οι οποίες θα είναι υπέρ όλου του τομέα και δεν έκανε καν μία συνεδρίαση με τους κοιόδης συγγητές, δεν άκουσε καμία πρόταση. Δεν είναι αλήθεια. Εμένα δεν με κάλεσε κανείς ε, εσά όλα όσα λέτε κυρία Ροντσούλη. Δεν είναι αλήθεια. Εμείς ζητήσαμε να κάνουμε συνεδριάσεις για να συζητήσουμε το έγγραφο και να κάνουμε συμβαστικές προτάσεις, αλλά εσύ δεν δέχτηκες. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, κυρία Πρόεδρε, ότι η έκθεση της κυρίας Ροντσούλη σε καμία περίπτωση δεν βελτιώνει τα δικαιώματα των ναυτικών και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη της τι είναι οι συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Είμαι απόλυτα απογοητευμένη και πραγματικά επαναλαμβάνω ότι αν πραγματικά πιστεύαμε σε κοινωνική Ευρώπη και αυτά δεν είναι προεκλογικές υποσχέσεις, δεν αφορά τι εκλογέ αυτό, είναι θέμα αρχή. Θέλουμε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά του. Αν πραγματικά πιστεύουμε σε αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα όσα έχουν υποβληθεί στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, όλα αυτά είναι η αίθουσα είναι πολύ πρακτική για την συνεδρία που κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ε, ποιοι θέλουν να μπουν στο κατάλογο μιλητών. Ψαρία σε Άγια. Άλλοι. Γιατί μετά θα κλείσει ο κατάλογος. Κύριε Ντεμπάκερ. Ο κύριος Ντεμπάκερ μετά. Και εγώ μετά. Εσείς μετά. με πνεύμα συμβασμού και διαπραγμάτευσης πάντα. Κυρία Μαρίσα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου, Θα φιλανδικά. Αν θέλετε μετάφραση, βάλτε τα ακουστικά, σας παρακαλώ. Λοιπόν, αν ε, η οδηγία για τις ε, επιχειρήσεις πώληση όπως ε, εφαρμοστεί εδώ όπως προτείνει η Επιτροπή, τότε σε αυτή την περίπτωση κατά την πώληση σκαφών από ένα κάτω μέλος σε άλλο προκαλούνται προβλήματα. Γιατί οι ναυτικοί θα ακολουθήσουν το σκάφος. Έτσι προτείνω αυτή η οδηγία να μην εφαρμοστεί τόσο εκτεταμένα όσο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτό θα μας οδηγούσε σε μια κατάσταση όπου τα σκάφη πολλούνται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μειώνεται το ρυθμό των θέσεων απασχόλησης. Νομίζω ότι οποιοδήποτε συμβιβασμό θα να περαιτέρω αυτή την πρόταση. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριληφθεί αυτή η οδηγία που ανέφερα, γιατί οδηγεί στην απώλεια θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, κάνω λάθος ε, στο ε, κουμπί. Δεν το έχω συνηθίσει. Λοιπόν, κύριος Ντεβάκερ. Δεν θέλω να προκαλέσω για καυγά, όχι, μόνο για να διευκρινίσω τη θέση μας. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε τόσο έντονε ε, συναισθηματικά συζητήσει, Εδώ πέρα ε, βασιζόμαστε σε δεδομένα που είναι πολύ σαφή για μένα τουλάχιστον. Γι' αυτό και συμφωνώ με την εισηγήτρια στην προσέγγισή τη, έχει υποβάλει τροπολογίε τι οποίε εμείς μπορούμε να στηρίξουμε γιατί βλέπουμε ότι και τα 28 κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία που προστατεύει ακριβώ την κατηγορία, την ειδική κατηγορία των ναυτικών. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, στην νομοθεσία Υπάρχει διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και οι ε, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων πολλές φορές έχουν ξεκαθαρίσει τις απόψεις τους για το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την υπόθεση η πρόταση τη Επιτροπή θα επιδεινώσει, θα δυσχεράνει την κατάσταση των ναυτικών σε πολλέ περιπτώσει. Γι' αυτό και η πρόταση τη εισηγήτρια ήταν να τροποποιήσουμε ε, σε πολλέ περιπτώσει, σε πολλά σημεία, την πρόταση τη Επιτροπή. Γι' αυτό και η ομάδα μου στήριξε αυτή την προσέγγιση, γι' αυτό καταλήγω σε αυτή την λίστα ψηφοφορία δεν χρειάζεται να ανάβουν τα αίματα. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει ε, σε αυτή την αίθουσα για το πώ θα επιλύσουμε το πρόβλημα. Έγινε η επιλογή των πολιτικών ομάδων. Έχετε λίστα ψηφοφορία. Παρακαλώ α μείνουμε ήρεμοι λοιπόν και α ψηφίσουμε. Πρόεδρο, νομίζω ότι όλοι άκουσαν το μήνυμα που θέλατε να απευθύνετε. Σρέντερ και μετά θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει η συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη. Έχω ένα πρόβλημα, διότι εδώ βλέπω μια υποστήριξη στην ιδέα οι τρύπε στο τυρί να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Έχουμε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο, διαθέτει κανόνες, κάθε εξαίρεση σημαίνει ότι υποσκάπτονται οι κανόνες. Τα είδαμε αυτά και στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων είδαμε πόσο δύσκολο είναι να ρυθμιστούν δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και ήταν σημαντική η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κλείσει κάποια παραθυράκια, κάποιες τρύπες στο τυρί. Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν καταρχήν καλό. Επέρχονται κάποιες βελτιώσεις, όμως βρίσκω ότι οι προτάσεις της συγγετρίας είναι εσφαλμένες και κάνουν, όπως είπα, τις τρυπε στο τυρί ακόμα μεγαλύτερες και δεν μπορεί αυτό να είναι που επιθυμούμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να απορρίψουμε τις τροποποιήσεις, τις, συγγνώμη, τις τροπολογίες της Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια πάλι και υπενθυμίζοντας ότι έχουμε βέβαια κάποια ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις συνθήκες ασφαλείας και εργασίας του προσωπικού των ναυτικών μεταφορών. Και αντιλαμβανόμαστε τις εθνικές ευαισθησίες. Θυμούμε και την τραγωδία του Κώστα Κονκόρδια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι εφοπλιστές κάνουν πραγματικά ό,τι μπορούν για να εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες ασφαλείας. Ωστόσο, θα σας δώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε την συζήτηση που συζήτηση πραγματικά δεν είναι, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε δεν υπάρχουν και θα περάσουμε στι τροπολογίε σα ευθύ αμέσω. Κυρία Εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω του συναδέλφου που κατάλαβαν τις προθέσει μου, τη γραμμή που θέλω να ακολουθήσω, αλλά επειδή άκουσα πολλά σλόγγαν σήμερα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η εξαίρεση δεν σημαίνει ότι τους προστατεύουμε. Ίσα ίσα, επειδή και τα 28 κράτη-μέλη έχουν ήδη νομοθεσία και ήδη προστατεύονται στη χώρα τους, για ποιο λόγο για κενά και ε, τρύπε στο τυρί, λυπάμαι κυρία Σρέντεν που τα λέτε αυτά, να επιμένουμε να αλλάξουμε μια οδηγία η οποία είναι παροχημένη και θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή, που εγγυάται πολύ περισσότερο και προ σου δίνει περισσότερη ασφάλεια. Όσον αφορά την ασφάλεια, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, αλλά ο καθένα θα πρέπει να αναφέρεται σε παραδείγματα τα οποία γνωρίζει. Και ειλικρινώ το παράδειγμα τη Κώστα Κονκόρδια δεν έχει καμία σχέση με την προστασία των ναυτικών. Δεν πρόκειται για μια περίπτωση στην οποία οι εφοπλιστέ δεν προστάτευσαν, πρόκειται για προσωπική ευθύνη και επειδή υπάρχει μια δικαστική διαδικασία πάρα πολύ σοβαρή εν εξέλιξη και ακόμα δεν έχει περατωθεί, θα ήθελα να σα ζητήσω να μην κάνετε παραδείγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την έκθεση αυτή. Οι εργαζόμενοι προστατεύονται. Υπάρχει μέρημνα για αυτού και επειδή αναφερθήκατε στην ασφάλεια, θα ήθελα να σα ε, καθησυχάσω. Η ασφάλεια για μένα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, γιατί προέρχομαι από ένα επάγγελμα ε, στο οποίο η ασφάλεια ήταν ε, πρωτίστη σημασία για του ασθενεί μου. Είναι δυνατόν να μην σκέφτομαι την ασφάλεια όταν είμαι υπεύθυνη για μια έκθεση η οποία κυρίως πρέπει να προτάσει την ασφάλεια και την ευημερία και πριν από τον εργοδότη και τον εφοπλιστή σε αυτή την περίπτωση. Είδα ότι σας αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιείτε διάφορα τσιτάτα και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι απορρίπτεται σε συγκεκριμένη ε, ε, νομοθεσία σήμερα θα αφήσετε τους εργαζομένους σπίτι τους διότι εάν απορρίψετε την ε, νομοθεσία και κάνετε αυτά τα οποία θέλετε θα αυξηθεί η ανεργία στους ναυτικούς. Εντάξει, ολοκληρώσαμε αυτή τη συζήτηση σε λίγα λεπτά θα έχουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, θα περάσουμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία μας. Έχουν όλα τα μέλη την κάρτα τους. Εντάξει. Θα περάσουμε λοιπόν ε, σε μια λευκή ψηφοφορία αρχικά για να είμαστε σίγουροι ότι ε, ψηφίζουμε όλοι καλά. Ένας φιλελεύθερος παραπάνω υπάρχει. Et parce que le est clos. Non, c'est pas clos. Bon, ça, πρόβλημα. Βάλτε καλά τις κάρτες σας. Έχουμε έναν φιλελεύθερο και έναν ΕΛΚ παραπάνω συντονιστές των φιλελευθέρων και του ΕΛΚ μπορούν ε, παρακαλώ να επιβάλλουν την τάξη. Α, δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Μπορείτε να αλλάξετε θέση. Alors, il faudrait que le groupe libéral mette de l'ordre οι φιλελεύθεροι θα πρέπει να βάλουν τάξη στις υποθέσεις τους. Και τώρα έχουμε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Ένα αναπληρωματικό μέλος λοιπόν θα πρέπει να φύγει. Δεν θέλω να επισέλθω στα της ομάδας σας, αλλά συνήθως τα αναπληρωματικά μέλη δημιουργούν το πρόβλημα. Εντάξει, Όλα εντάξει λοιπόν. Δεν κινείται κανένας. Να ψηφίσουμε. Περνάμε στο σημείο 6. Για την σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση για την υιοθέτηση ε, της οδηγίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου minimum για τις ελάχιστες ε, ελάχιστους όρους για την αύξηση της γενετικότητας των εργαζομένων μεταξύ των μελών, αυξάνοντας ε, ε, την εφαρμογή των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Η κυρία Ρέτεν ήταν η συγγήτρια. Λοιπόν, για αυτή τη ψηφοφορία δεν θα ισχύει για τις υπόλοιπες. Για πρώτη φορά θα εφαρμόσουμε τον νέο μας ε, κανόνα 195.3. Δηλαδή ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ε, και πλέον μιλάμε για ονομαστική ψηφοφορία. Υπερθυμίζω το πνεύμα του κανόνα. Η ψηφοφορία γίνεται ονομαστική όταν έχουμε την τελική ψηφοφορία για ε, έκθεση πρωτοβουλίας ή τελική ψηφοφορία για νομοθετική έκθεση. Μόνο όμως ε, στον καθορισμό της εντολής. Δηλαδή στο τέλο ε, τριμερού διαλόγου διαπραγμάτευση δεν πρόκειται για ονομαστική ψηφορία. Εδώ πέρα μιλάμε για την τελική έγκριση τη έκθεση Ρέτεν σε δεύτερη ανάγνωση για την βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων πνευματική δεξιοδότησης. Νομίζω ότι ήμουν σαφής στις εξηγήσεις μου. Θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Έναρξη λοιπόν. Έχουμε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ και από την Άλντα. C'est bon ou pas Il faudrait de l'ordre au sein du PPE. Λύστε το πρόβλημα παρακαλώ στο ΕΛΚ και στην ΑΛΔΕ. Est-ce que tous les libéraux peuvent lever la main? Μπορούν να σηκώσουν το χέρι τους τα μέλη ε, των φιλελευθέρων.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 Εντάξει, λοιπόν, έχει επιβληθεί η τάξη στις γραμμές της ΑΛΔΕ και του ΕΛΚ. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Σαράντα υπέρ, μία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και στο σύνολο της ομάδας διαπραγμάτευσης. Ε, Σημείο 7. Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με του ναυτικού που τροποποιεί τι οδηγίε 2008-94 2009-38, 2002-14, 98-59 και 2023. Έκθεση της κυρίας Ροτζούλη. Για τον ε, τίτλο έχουμε τρεις ε, τροπολογίες που σφίζουμε από κοινού, Ένα, 12 και 11 και 12 της εισηγήτριας για να διαγραφεί ε, ο τίτλος του άρθρου 5 και του άρθρου 6 της πρότασης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Tout le monde a pu voter. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 18 υπέρ, 23 κατά, 3 αποχές, απορρίπτεται. Σχόλια εκτό μικροφώνου. Λέει πρόεδρο δεν «Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Υπάρχει μια θέση εκεί κάτω, βλέπω. Για τα άρθρα. Άρθρο 1, παράγραφος 1α, τροπολογία 20, υπέρ κατά, αποχές, επαλήθευση για την τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. 22 Σρέντερ για τη διαγραφή του άρθρου 1 παράγραφος Παράγραφος 3. Το άρθρο υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ζητώ συγγνώμη, απλώς δεν είναι εύκολο Θα αυτήν την αίθουσα να δούμε ποιοι έχουν ψηφίσει. Πέρας. 19 ψήφοι υπέρ, 23 κατά, 3 αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 2, σημείο 1. Άρθρος 1, παράγραφος 7 αντίστοιχη. Τροπολογία 7 του εισηγήτρες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Κλοντέτ Αβέλα Μπαλτατσίνο. Για διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας δούμε. Άρχεται. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 22 υπέρ, 23 κατά. Μηδέν αποχές. Απορρίπτεται. Για το ίδιο σημείο, τροπολογία 23, Σρέντερ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Τροπολογία 8 εισηγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Tout monde a pu voter, le vote est clos. Πέρας. 18 υπέρ, 25 κατά, 2 αποχές, πράγματι απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Της υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Α, 24 διορθώνει η πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 24. Tout le monde Πέρας. 24 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν 24. Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο 2, τροπολογία 27. Δεν ξέρω νου. 27 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 27. Tout le monde a pu voter, le vote Πέρας ψηφοφορίας, 22 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Ελίζαμπετ Σρέντερ. Τροπολογία διαγραφής ταυτόσιμη με την 29 της ε, Μπαλτατσίνο. της ψηφίσουμε λοιπόν από κοινού υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτονται οι δύο αυτές τροπολογίες. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στα εκτιμώντας. Εκτιμώντας 2. Η 2 δεν έχει αντικείμενο, όπως και η 5, 6. Περνάμε λοιπόν στο εκτιμώντας 1. Τροπολογία 13, Σρέντερ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote... 22 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται 13. Στο 5. Τροπολογία 3 εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 14. τη Βελτατσίνο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στο 7. Τροπολογία 4 ηγητρία. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. Εκτιμώντα 10. Τροπολογία 15. Η οποία απεσύρθη. Περνάμε λοιπόν στην 11. Αντιορθώνει προέδρο. Τροπολογία 16 τη Μπαλτατσίνου. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 17 της ίδιας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 της ίδιας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 της ίδιας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε από του συνόλου της έκθεσης. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται. Le vote est Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 14 υπέρ, 22 κατά, 9 αποχές. Θέλετε να παρεμβείτε, η συγγήτρια, πριν από την ε, ψηφοφορία για την νομοθετική πρόταση. Που δεν θα γίνει αυτή η ψηφοφορία γιατί απερίφθη η έκθεση. Ευχαριστώ. Δεν θα υπάρξει λοιπόν θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το κείμενο. Και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία θα δούμε αν η Επιτροπή θα επιβεβαιώσει την πρότασή της όπως ε, αυτή είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Στο σημείο 8 περνάμε στα συμπεράσματα της ε, διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο για την ε, 96-71 ε, για, για την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχή υπηρεσιών. Euh, Ωραία. Θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία για το κείμενο όπως έχει εγκριθεί από τη διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το επιβεβαίωσε και η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων στις 26 Φεβρουαρίου του 2014 και επιβεβαιώθηκε στην Κορεπέρ τη 5 η Μαρτίου 2014. Άρχεται η ψηφοφορία, δεν είναι ονομαστική κλίση. Έχουμε έναν φιλελεύθερο επιπλέον. Έναν ε, φιλελεύθερο και έναν από το ΕΛΚ επιπλέον έχουμε. Les choses sont en ordre. Ωραία. Ρυθμίστηκαν όλα. Και πέρασε η ψηφοφορία. 30 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και τη διαπραγματευτική ομάδα. Πριν περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία, ίσως πρέπει οι φιλελεύθεροι να προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν λίγο τι γίνεται. Φαίνεται να υπάρχει ε, μία σύγχυση. φαίνεται σαν να έχουν οι φιλελεύθεροι μία θέση λιγότερη, διότι ε, είχαμε ένα μέλος ε, το οποίο έφυγε και πήγε στους σοσιαλιστές και δεν μπόρεσε να υπάρξει ολομέλεια για να ρυθμίσει. Ε, επομένως έχουμε πέντε μέλη και όχι έξι πλέον ε, στην ομάδα. Πάμε στο σημείο 9 και θα ψηφίσουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένσταση για την ε, έκθεση της Προ... Επιτροπής που ρυθμίζει τον κανονισμό 233 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ε, Ταμείο Βοήθειας στους ε, πιο ευάλωτους. Θέλουμε να ψηφίσουμε τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, οι οποίες θα επιτρέψουν την εφαρμογή ε, του Ταμείου για τους πιο ευάλωτους για την επόμενη οικονομική περίοδο. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, χωρίς ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter. Le τη ψηφοφορία. 44 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Αποφασίστηκε λοιπόν το ζήτημα. Στο σημείο 10 ψηφίζουμε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για αίτημα το οποίο σχετίζεται με την επιχείρηση VDC Technology στην Ιταλία, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 11. Κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην ε, ε, Παγκοσμιοποίηση. Έτοιμα της ομάδος Σαντάνα στην Ισπανία. Του ομίλου Σαντάνα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η ψηφοφορία και θα ήθελα να ζητήσω σε όσους ε, πρέπει να φύγουν από την αίθουσα να φύγουν ησύχως το συντομότερο δυνατόν.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε, διότι έχουμε ένα νέο σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 12 θα Έχουμε την ακρόαση της κυρίας Μαντλίν Σέρμπεν που είναι υποψήφια για νέα θητεία ως εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την κατάρτιση. Ο οργανισμός ε, ETF που εδρεύει στο Τωρίνο. Η κυρία Σέρμπαν επελέγει από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Απριλίου του 2009 για εκτελεστική διευθύντρια από 1η Ιουλίου του 2009 του Ιδρύματος και ε, στο τέλος της θητείας της αυτή των 5 ετών ε, στις 30 Ιουνίου του 2013 προτάθηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2013 να ανανεωθεί η θητεία της ε, κυρίας Σέρμπαν και εγώ ενημερώθηκα από την για την απόφαση αυτή από μια επιστολή του ε, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου. δεν είχαν ενημερωθεί τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης. Απάντησα αμέσω ε, και ανέφερα την έκπληξή μου για το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε η Επιτροπή Απασχόλησης για αυτή τη διαδικασία, διότι το άρθρο 10 του κανονισμού του οργανισμού προβλέπει ότι η εκτελεστική ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί να κληθεί ε, για ακρόαση και παρουσία ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να απαντήσει και σε ερωτήσεις ε, των μελών. Έχω λοιπόν τη μεγάλη τιμή να υποδεχθώ εδώ την κυρία Σερμπάν, την οποία γνωρίζουμε, είναι γνωσμένου κύρους, άσκησε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντά της στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά περίπου και κατόπιν τα μέλη της Επιτροπής μας θα σας θέσουν ερωτήσεις και ε, θα έχουμε μια διαδικασία ερωταποκρίσεων ε, κατά τα συνήθη κάθε φορά που έχουμε ακρόαση ε, για ανάληψη καθηκόντων γίνεται κάτι αντίστοιχο. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερως για την πρόσκληση ε, την οποία όπως σας είπα αποδέχομαι τα τιμή. Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την ε, πολύ μεγάλη υποστήριξη ε, στη διάρκεια της πρώτης μου θητείας ως εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού ε, και πρέπει να πω ότι αν υπήρξαν αποτελέσματα από πλευράς του οργανισμού αυτό συνέβη διότι υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο είναι και το πιο σημαντικό όπως πάντα αναφέρω. Με την άδειά σας τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες για την επόμενη θητεία εάν συμφωνήσετε να αναλάβω καθήκοντα από 1η ε, Ιουλίου του 2014 και θα σας τα παρουσιάσω αυτά στην Αγγλική. Όπως θα γνωρίζετε, από τότε που είχα έρθει ε, σε όλες τις πέντε ετήσιες ακροάσεις που γίνονται στην αρχή κάθε έτους για να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες του ETF και να σας παρουσιάσω και τις ε, ιδέες μας για το μέλλον των δραστηριοτήτων μας, ε, το ε, Ίδρυμά μας της επαγγελματικής εκπαίδευσης ε, ενδιαφέρεται για την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 συντάξαμε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική 2014-2017. Εάν λοιπόν μου επιτρέψετε να συνεχίσω τη θητεία μου ως εκτελεστική διευθύντρια θα διασφαλίσω ότι όλοι οι στρατηγικοί στόχοι και οι δραστηριότητες προσανατολισμού που αναφέρονται στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές 2014-2017 θα εφαρμοστούν. Με την άδειά σα ε, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στους στρατηγικούς στόχους ε, όπως έχουν εγκριθεί. Καταρχάς λοιπόν αναφερόμαστε στην ενίσχυση των πολιτικών που βασίζονται σε απτά στοιχεία και σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε στην ανάλυση πολιτικής καταρχάς και θα ήθελα να σας αναφέρω ότι στην περίπτωση της ανάλυσης πολιτικής αναφερόμαστε σε μια ε, ανάλυση συστημική αλλά και με θεματικές ενότητες. Ο βασικός στόχος για το 2014-2014 είναι ο εξυγχρονισμός των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ε, με τη διαβίου μάθηση και ο δεύτερος στόχος είναι η αύξηση των διατάξεων για την επαγγελματική κατάρτιση στα ε, πλαίσια της αγοράς και της κοινωνικής συνοχής. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι το Ίδρυμά μας είναι ο μόνος ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος ε, δρά στην ε, παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη. Δρούμε λοιπόν προσπαθώντας να προσδώσουμε ζωή και να ε, υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής της εξωτερικής διάστασης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και να ε, υπάρχει μεγάλη σημασία και στην αγορά αυτών των δράσεων. Δρούμε λοιπόν αποκλειστικά εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς το παρόν δραστηριοποιούμεθα σε 47 ε, ε, χώρες που ανήκουν στην περιοχή διεύρυνσης, αναφέρομαι στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Τουρκία και σε χώρες οι οποίες υποστηρίζονται από την πολιτική γειτονία και εδώ αναφέρομαι στην Ανατολική και Νότια Μεσόγειο, καθώς επίσης και την Ανατολική Ευρώπη και επιπλέον ε, συνεργαζόμαστε και με την Κεντρική Ασία στον τομέα της ανάπτυξης ε, και συνεργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι ασχολούμαστε με την εξωτερική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά στα πλαίσια των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ε, μία γέφυρα διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και αυτών των χωρών ε, και δεν εξετάζουμε αποκλειστικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά προσπαθούμε να... Ε, συνεργαστούν τα κράτη-μέλη με χώρες ε, των ενδιαφερόντων τους και ε, συγκεκριμένων δράσεων. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε τι κάνουμε και πώς διαχειριζόμαστε αυτούς τους στρατηγικούς στόχους ε, είναι αντικείμενο μιας πολιτικής ανάλυσης η οποία γίνεται κάθε δύο χρόνια με τις χώρες εταίρους ε, η οποία καλείται διαδικασία του Τωρίνο και έχει ε, πηγή έμπνευση στη διαδικασία της Κοπενχάγης που ξεκίνησε στα κράτη-μέλη το 2002 και με τη βάση όλων των αναγκών που έχουν οι χώρες αυτές για την ενίσχυση των πολιτικών για τους ανθρωπίνους ε, πόρους επιλέγουμε κάποιους θεματικούς στόχους να σας υπενθυμίσω ότι το Ίδρυμά μας έχει ως αποστολή να διασφαλίσει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών και ε, μέσω ανταγωνιστικότητας και μέσω κοινωνικής συνοχής ε, για τις χώρες αυτές. Συνεπώς, κάθε φορά που αναφερόμαστε στην κοινωνική συνοχή και στην ανταγωνιστικότητα, ε, θεωρούμε ότι πρόκειται για εγκιάρσιους τομείς δράσης, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες θεματικές ενότητες οι οποίες αναφέρονται στα προσόντα και στα ε, συστήματα ε, πιστοποίησης των επαγγελματικών ε, προσόντων, διακυβέρνηση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, απασχόληση και αποσχολησιμότητα. Ένας άλλος θεματικός τομέας είναι οι δεξιότητες και η μετανάστευση και ένας τελευταίος ε, στόχος, τον οποίο θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη ε, ε, σας, είναι επιχειρηματικό γίγνεσθε. Έτσι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας, αλλά φυσικά όλα αυτά θα είναι δυνατά μόνο εάν ο οργανισμός διαθέτει τους μηχανισμούς και τα εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να επιτύχουμε τους ποσοτικούς στόχους όπως ε, τους έχουμε καθορίσει, αλλά να υπάρχουν και ποιοτικοί στόχοι. Με άλλα λόγια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν κάποιες συνέπειες οι δράσεις μας. Και για την επόμενη θητεία θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ενισχύσουμε την αλλαγή της διαφορετικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες αυτές τις χώρες εταίρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε ποιες είναι οι ανάγκες πολιτικές των χωρών αυτών, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει στη συνέχεια να συνάδει με τη στήριξη μέσω των διαφόρων μέσων που θα δοθεί ε, στις διάφορες χώρες και να δίνεται στις χώρες αυτές της διεύρυνσης, της προενταξιακής διαδικασίας, ε, της ανατολικής συνεργασίας ε, και της πολιτικής γειτονίας. Να σας υπενθυμίσω και τα σημεία 30-39 του 2008 που λένε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει συνέχεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ του έργου του οργανισμού και άλλων ε, δραστηριοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο παροχής ε, συνδρομής στις χώρες αυτές. Από μόνοι μας φυσικά δεν μπορούμε να επιτύχουμε και πάρα πολλά, γι' αυτό συνεργαζόμαστε ε, με ε, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού και φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτό το διαρθρωτικό διάλογο ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει τις διάφορες ε, Γενικές Διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Εξωτερική Υπηρεσία Δράσης για να δούμε τι είναι καλύτερο για τις χώρες αυτές και τι ακριβώς κάνουν οι άλλες Γενικές Διευθύνσεις, η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης και ΔΕΦΚΟ θα διασφαλίσουν στη διάρκεια του προγραμματισμού η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ δεν δρά μόνο άμεσα στις χώρες αυτές, αλλά ε, μεγάλο ποσοστό είναι τμήμα του προγραμματισμού που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να υπάρχουν προτάσεις για τα οποία, ε, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό. Και εδώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ των όσων θεωρούμε ε, ως... Ε, Συμβουλές πολιτικές, δημιουργία δυνατοτήτων, δικτύωση μεταξύ των κρατών μελών και των χωρών εταίρων και το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα κονδύλια. Όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, ελπίζω ότι ο οργανισμός μας θα συνεχίσει να, λαμβά... να έχει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που είχε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μπορεί να δεσμεύσει και να δαπανίσει καταλήλως τις πιστώσεις υποχρεώσεων και όχι μο... τις δεσμεύσεις, συγγνώμη, αλλά ε, και με καλά αποτελέσματα όπως φαίνεται και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, για την καλή χρήση των πόρων αυτών, βελτιστοποιώντας το στο, μέτρο του δυνατού και φροντίζοντας να έχουμε ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε και τις ε, συστάσεις στην, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου κάθε φορά που έρχονται να μας επισκεφθούν, ε, αλλά πρέπει να πω ότι από τις επισκέψεις που είχαμε οι συστάσεις τους δεν μπορούν να αμφισβητήσουν ε, τη δυνατότητα που έχει ο οργανισμός να διαχειρίζεται καταλήλως τους πόρους τους. Είμαι ιδιαίτερα καθησυχασμένη λοιπόν που ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους ε, στρατηγικούς στόχους ε, ε, της διαδικασίας της ενδιάμεσης που μόλις ξεκίνησε το 2014 και ελπίζω ότι επειδή ο οργανισμός είναι τόσο σημαντικός δεδομένου ότι είναι και ο μόνος ο οποίος ε, δρά σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους όπως ε, ε, συμβαίνει τώρα και να μην υπάρξουν γραμμικές περικοπές, αλλά να γίνει πρώτα ανάλυση των προτεραιοτήτων και για τα επόμενα χρόνια. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Για την επόμενη θητεία θα ήθελα να προτείνω αυτά λοιπόν και είμαι στη διάθεσή σας σε περίπτωση που θέλετε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup euh, de cet euh, exposé très, très exhaustif euh, de Ευχαριστούμε για αυτή την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη εισαγωγή. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μαγαζατιέ μετά Θέρκας. προ το παρόν οι δύο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά εκ μέρου ε, του ΕΛΚ να ευχαριστήσω την κυρία Σερμάν για αυτή την ε, ιδιαίτερα σαφή και ολοκληρωμένη εισαγωγή σε ό,τι φορά το έργο που έχει επιτελέσει τα τελευταία πέντε έτη αλλά και για τα όσα ακόμα μένουν να γίνουν Γνωρίζοντα βεβαίω, όλοι το γνωρίζουμε, ότι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική Εκπαίδευση έχει θεμελιώδη ρόλο να διαδραματίσει σε μια χρονική συγκυρία που η ενεργεία αποτελεί το πρωταρχικό σημείο προβληματισμού σε όλα τα κράτη-μέλη και βλέπετε αυτή τη διάκριση μεταξύ της πολιτικής γειτονίας και της προσχώρησης κάποιων κρατών αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και θα ήθελα, κυρία, να ξεκινήσω από τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ε, ξεκάθαρα στοιχεία, εύρωστα στοιχεία, που είναι πολύ δύσκολο να τα βρούμε, γιατί οι αναλύσεις ε, που κάνατε για το 2014 δεν είναι ίδια ίδιες για το 2009. Τροποποιείται λοιπόν η κατάσταση. Η κύρια δυσκολία, και εδώ θα ήθελα να επικεντρωθώ, πώς θεωρείτε ότι μπορείτε να παρέμβετε εσείς ό,τι αφορά την επιτάχυνση της αντίδρασης. Η αντίδρασή μας σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα της ε, εκπαίδευσης, ε, τις ανάγκες που μεταβάλλονται και επιταχύνονται στον τομέα των επιχειρήσεων αφενός, αλλά και των εργαζομένων από την άλλη. Για μένα είναι απολύτως κυριαρχική σημασία αυτό το θέμα, γιατί μπορούμε να έχουμε καλές ιδέες, καλές προοπτικές, όμως ε, το πρόβλημα του χρόνου η χρονική διάσταση για την ανταπόκρισή μας ε, στο ζήτημα της ανεργίας είναι πολύ σημαντικό. Ο χρόνος της κατάρτισης δεν είναι ο ίδιος με το χρόνο της επιχείρησης. Αυτό είναι το πρώτο πεδίο στο οποίο θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη. Δεύτερο σημείο. Πώς εξελίσσονται και οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις ε, αυξημένες ε, απαιτήσεις ε, της απασχόλησης στην Ευρώπη εφόσον σήμερα όλες οι προοπτικές το 2020, για την Ευρώπη 2020, βλέπουν ότι υπάρχει σημαντική μεταβολή του πεδίου στο κάτω μέρος της πυραμίδας ε, χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο αριθμό με λιγότερες δεξιότητες και στο πάνω μέρος της πυραμίδας χρειαζόμαστε λιγότερους εργαζομένους με περισσότερες δεξιότητες. Επομένως, έχουμε αυτή την μεταβολή ε, των δεξι... της ε, κατεύθυνσης των δεξιοτήτων προς την κορυφή της πυραμίδας. Επομένως, πάντα θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Τρίτο σημείο. Πώς μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά την κατανομή αυτών των προτεραιοτήτων που αναφέρατε σε όλα τα κρατημέλη. Πώς ακριβώς θα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε, από τις δικές σας αναλύσεις, όλα τα στοιχεία, τα στατιστικά που συλλέγονται, πώς όλα αυτά μεταφράζονται στην πράξη. Γιατί και εδώ πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, κατά τη γνώμη μου. Τέλος, και τελευταία μου ερώτηση, μιλήσατε για ε, την ε, κύρωση του κεκτημένου. Αυτά μας απασχολούν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι δεν είμαστε αρκετά ταχείς και αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά αυτή την κύρωση των κεκτημένων. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να το δούμε πιο πρακτικά. Θεωρείτε ότι αυτό ισχύει γιατί ακολουθήσαμε μια πλέον ε, ακαδημαϊκή προσέγγιση πέραν του δέοντος. Όμως ε, σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ καλό εργαλείο που όμως ε, δεν μας δίνει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Ιδίως αναφέρομαι σε κοινωνικές ομάδες ε, που επλήγησαν ιδιαίτερως από την κρίση. Συγκεκριμένα αναφέρομαι για παράδειγμα στις γυναίκες που έχουμε και άλλες ομάδες ε, εργαζομένων και το καθεξής. Σε αυτά τα τέσσερα σημεία λοιπόν θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο. Κυρία Σέρμπαν. Σας ευχαριστώ πρώτα για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου για τις ε, χώρες μέλη. Θα αναφερθώ όμως στις εμπειρίες που έχουμε στις χώρες εταίρους και που σίγουρα δεν είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι συμβαίνει σε ορισμένες από τις χώρες μέλη. Ορισμένες από τις σκέψεις μου πιστεύω ότι ισχύουν και για τις χώρες μέλη. Όταν αναφερόμαστε στην ανεργία και σε λύσεις βασισμένες στα στοιχεία, evidence-based δηλαδή, πρώτα βέβαια πρέπει να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και πώς θα καθορίσουμε τις διάφορες παραμέτρους. Όπως είπατε κι εσείς, και τα συζητούμε βέβαια τα στοιχεία αυτά, πρώτα-πρώτα είναι το στοιχείο του χρόνου. Εφόσον βρούμε στο επίπεδο πολιτικών και συστημάτων, η αλλαγή συστήματος χρειάζεται χρόνο. Και δυστυχώς η ανεργία είναι σήμερα και θίγει τους ανθρώπους σήμερα. Έτσι σε όλες τις δράσεις που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε στις χώρες μέλη, κοιτούμε πρώτα-πρώτα να βρούμε μια γρήγορη λύση, quick fix ταυτόχρονα όμως επεξεργαζόμαστε και το ίδιο το σύστημα. Γιατί είναι πιο σημαντικό να δρά κανείς προληπτικά παρά θεραπευτικά, δηλαδή για να διορθώσει τα όσα προκαλεί το σύστημα, για παράδειγμα ε, δυσκολίες συνέχειας. Και για τις ταχύες λύσεις, και δεν θα πω βέβαια για μακροπρόθεσμες, μάλλον μεσοπρόθεσμες δράσεις, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δεν υφίσταται πραγματικός διάλογος ανάμεσα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην επιχείρηση. Και δυστυχώς, εδώ και χρόνια μιλούμε για αυτά, αλλά ακόμη δεν είναι όλοι διαθέσιμοι και έτοιμοι και από τις δύο πλευρές να συμμετάσχουν. Έχουμε πολλές καλές εμπειρίες και σημαντικό αριθμό καλών πρακτικών που όμως δεν έχουν λάβει χαρακτήρα συστηματικό. Και γι' αυτό απλώς είναι τυχαία σύμπτωση όταν πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας μπορούν να υποφεληθούν εν τέλει από όλα αυτά. Από τη μια μεριά λοιπόν αυτά διότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και δεν μιλώ μοναχά για την επίσημη εκπαίδευση αλλά και για την επίσημη. είναι πολύ άκαμπτος ο κόσμος αυτός και συντηρητικός και αυτό διότι τους λείπει η πληροφορία και η γνώση για το πώς να δράσουν αναφέρομαι πάλι στις χώρες εταίρους του ETF. Εφόσον αναφέρομαι σε αυτό, στη δυσκολία της αλλαγής, είναι διότι γίνεται πολύ λίγη επένδυση σε δασκάλους και σε εκπαίδευση εκπαιδευτών. Σε εκπαιδευτές δηλαδή και σε εκπαίδευση εκπαιδευτών. Διότι η δουλειά τους δεν αξιολογείται από την κοινωνία. Από τη μια μεριά λοιπόν δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητο ότι οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Και από την άλλη μεριά είναι ο κόσμος των επιχειρήσεων. Δυστυχώς πολλές από τις επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα στην φάση του προβληματισμού ή της σκέψης τους ότι είναι μέρος της φιλανθρωπίας να καθίσουν να συνεργαστούν με την εκπαίδευση. Το μήνυμα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις είναι ότι δεν είναι φιλανθρωπία εκ μέρους τους. Είναι υποχρεωσή τους να διασφαλίσουν ότι θα μπουν σε διάλογο με όλη αυτή τη δουλειά και να καταθέσουν και αυτά που θεωρούν ότι είναι τμήμα της λύσης. Το world-based learning, για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μάθεις, να εκπαιδευτείς δίθεν μέσα σε ένα ελεφάντινο πύργο και ξαφνικά να θεωρήσεις ότι μπορείς να βγεις στην αγορά εργασίας. Επίσης, θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ενισχυθούν. Διότι αυτά τα μέτρα λιτότητας δεν επιτρέπουν να προχωρήσετε. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη υποστήριξη από αυτήν την άποψη. Αυτά νομίζω ε, ότι είναι τα σημαντικά. Δηλαδή ο χρονισμός των δράσεων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δηλαδή πρέπει να κάνουν περισσότερα για να φροντίσουν να συμμετάσχουν περισσότερο. Τώρα οι απασχολούμενοι έχουν τέλος πάντων τα προσόντα που διαθέτουν και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια προσόντα διαθέτουν. Δυστυχώς στις χώρες, χώρες εταίρους τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφανείς ό,τι αφορά τα προσόντα των ε, προσώπων αυτών, διότι υπάρχουν και τίτλοι και διπλώματα τα οποία δεν εκδίδονται με διαφανή τρόπο και γι' αυτό οι δεξιότητες που απαιτούνται ίσως να μην είναι οι ε, σωστές, δηλαδή οι δεξιότητες που διαθέτουν ίσως να μην είναι αυτές που απαιτούν οι νέες συνθήκες εργασίας και οι νέες τεχνολογίες. Είναι πολύ δύσκολο όμως επειδή δεν γνωρίζουμε τι διαθέτουν να δούμε και να σχεδιάσουμε την κάλυψη των αναγκών. Πρέπει λοιπόν οι χώρε εταίροι να καταστήσουν διαφανή τα, τις δεξιότητες αυτές και διαφανείς. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην πρώτη σας ερώτηση για την αξιολόγηση της πρώτερης εκπαίδευσης, του prior learning, πρώτης, πρώτερης μάθησης. Να δούμε δηλαδή οι απασχολούμενοι τι δεξιότητες διαθέτουν και είτε εφόσον αυτά έχουν ε, αποκτηθεί μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης ή και στη δουλειά. Τώρα πού βρίσκεται η δυσκολία σε αυτά. Στις χώρες εταίρους η δυσκολία προκύπτει από την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας των μηχανισμών. Υπάρχει δε μέγας κίνδυνος απότομης όθησης της έκδοσης των προσόντων εφόσον δεν υπάρχει η διασφάλιση της ποιότητας. Αυτό είναι το, ε, το ενδεχόμενο διαστρεβλωμένο αποτέλεσμα των μηχανισμών αυτών. Εκδίδονται δηλαδή πτυχία προσόντων που δεν είναι όμως εξασφαλισμένη η ποιότητα. Δηλαδή δημιουργούμε προσδοκίες που ωστόσο δεν ανταποκρίνονται ποτέ στις ε, προσδοκίες των αντίστοιχων αγορών. Ονειροπολώ τώρα βέβαια ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή που θα έχουν όλες οι ε, χώρες μέλη μια συντονισμένη ενέργεια. Πιστεύω όμως ότι το ευρωπαϊκό project αποτελεί την λύση για, τον, ε, για την Ήπειρο. Και ελπίζω πραγματικά ο συντονισμός αυτός θα μπορέσει να συνεχιστεί και ε, η συνέργεια θα επιτύχει, η Ευρώπη θα μπορέσει να μιλήσει με μια φωνή και οφείλω να πω ότι για μας είναι πολύ καθαρό πόσο απαραίτητο είναι αυτό και κυρίως όταν βρούμε σε χώρες όπως η Ουκρανία που εδώ είναι καυτό θέμα ε, τις μέρες αυτές σε χώρες όπως οι αραβικές χώρες όπου όλοι χρειάζονται περισσότερη Ευρώπη και αυτό το τονίζω χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη σε περισσότερη ευρωπαϊκή παρουσία σε όλες αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρκας. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Σερβάν, θα ήθελα εξ ονόμαστος των Σοσιαλιστών Ευρωβουλευτών, εν συντομία καταρχάς να αναγνωρίσω το έργο σας και τα όσα κάνατε εσείς στο Ίδρυμά σας και να σας υποστηρίξω ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε αίσιο τέλος η στρατηγική η οποία έχετε χαράξει μέχρι το 2020 και αυτό το ενδιάμεσο στάδιο μέχρι το 2014. 17, συγγνώμη, διορθώνει ο Και να σας πω ότι εμείς πραγματικά θα ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι αν συνεχίσετε αυτό το έργο. Εμείς οι σοσιαλιστές είμαστε συντηρητικοί. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει ε, να μην αλλάζουμε ό,τι δεν λειτουργεί, αλλά πρέπει σίγουρα να διατηρούμε αυτό το οποίο έχει αποτέλεσμα. Ζούμε κάποιες στιγμές οι οποίες ε, προφανώς ε, για όποιον έχει ανοιχτά τα μάτια του είναι πολύ σημαντικές για την Ευρώπη και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το μέλλον όλων των εταίρων μας, ε, όλων όσων βρίσκονται εκτός των συνόρων μας και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς το μέλλον μας εξαρτάται και από το μέλλον τους. Και αν δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς, ε, απειλείται το δικό μας το μέλλον. Και αυτή η αλληλεξάρτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει ίσως ε, το ευρωπαϊκό σήμα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προέχει στην Αραβική Άνοιξη και στην Άνοιξη οποιασδήποτε χώρας. Δεν αξίζει να γίνονται απλώ διπλωματικές προσπάθειες σε θέματα ε, εξωτερικής πολιτικής, ε, ε, σε θέματα παιδεία, σε θέματα οποιοδήποτε θέμα, εάν είναι διαιρεμένες 28 πολιτικές και πρέπει να έχουμε αυτή την εξωτερική διάσταση η οποία θα παρουσιάζει την Ευρώπη για αυτό που είναι μια ενδιάμεση δύναμη ίσως σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία όμως έχει τη φιλοδοξία να προτείνει στον κόσμο και να είναι μια ήπια δύναμη, αλλά θέλουμε να είμαστε δύναμοι, διότι έχουμε πράγματα να πούμε και ε, θέλουμε να θριαμβεύσει το μοντέλο, το μοντέλο μας. Και εσείς φυσικά συνεισφέρετε πολύ σημαντικά. Το να δίνουμε δυνατότητες στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε κατάρτιση είναι ε, η πρακτική εφαρμογή του μοντέλου μας μπορεί να μην έχει θεαματικά αποτελέσματα, αλλά ε, είναι μια προληπτική πολιτική και πολύ καλύτερα να προλαμβάνουμε τις συγκρούσεις από το να πρέπει να τις ε, ε σταματήσουμε στη συνέχεια. Και ίσως ε, οι πιο προσεκτικοί παρατηρητές να βλέπουν ότι οι συγκρούσεις έχουν σχέση και με την έλλειψη ελπίδας για το μέλλον, έλλειψη αξιοπρέπειας του ατόμου, έλλειψη εργασίας, έλλειψη ποιότητας στην εργασία και απελπισία. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι και η απελπισία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ε, παθολογικές απαντήσεις. Εσείς λοιπόν ε, κάνετε ένα πολύ σημαντικό έργο και για αυτούς αλλά και για μας. Θα ήθελα λοιπόν αναγνωρίζοντας το έργο σας, να υπενθυμίσω ότι δεν ε, είναι κίνητρο μόνο η γενοδορία για τη συνεργασία. Έχει διπλή χρήση αυτή η συνεργασία. Η Ευρώπη διδάσκοντας μαθαίνει κιόλα. Και θα ήθελα να σας θέσω και μία ερώτηση. Ε, μαθαίνει διότι δυστυχώς Βλέπουμε ήδη και στους δρόμους ε, και στην Ευρώπη, ε, στην Ελλάδα για παράδειγμα, ανθρώπους που τους έχει πλήξει η κρίση. Βλέπουμε μια κοινωνία η οποία πολύ μοιάζει με τις αναθεώμενες χώρες. Ε, βλέπουμε ε, πολύ μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης, ε, ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν χάσει θέση εργασίας, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το σχολείο και χάνουμε ένα πολύ σημαντικό εργατικό δυναμικό και αυτό φυσικά δεν διαφέρει και πολύ από το εργατικό δυναμικό που βλέπουμε στην Τουρκία ή και σε αναδυόμενες χώρες. Θεωρώ λοιπόν ότι η μέθοδό σας και η απόπειρα η οποία κάνετε, και εδώ έρχεται και η ερώτησή μας, πώς θα μπορούσε να ανακυκλωθεί σε αυτή την ε, ε, λιγότερο ευνοημένη Ευρώπη που υπάρχει, διότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Γερμανία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Ευρώπη είναι οι άνεργοι της Αθήνας, οι καταστρεμμένες επιχειρήσεις της Πορτογαλίας, άνθρωποι που έχουν χάσει την κλωστοεφαντουργία τις θέσεις εργασίας τους και δεν έχουν άλλες δεξιότητες. Θα μπορούσατε ίσως και εσείς να προσέξετε αυτή την εσωτερική ε, δημιουργία ενός τρίτου κόσμου που δυστυχώς ε, δημιουργείται στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να τον υποστηρίξουμε. Και επίσης να υποστηρίξουμε και κάτι ακόμα και με αυτό ολοκληρώνω, το οποίο είπατε και το λησμονούμε εδώ στην Ευρώπη. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι ή θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, συνδικάτων ε, και πολύ καλός κοινωνικός διάλογος, ιδάλλως η θα υπαρχει στενη συνεργασια μεταξυ επιχειρησεων συνδικατων και πολυ καλος κοινωνικος διαλογος δαλωση η καταρτιση και η εκπαίδευση είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Σα Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω, ε, ο μόνος τρόπος να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η συνεργασία μας. Πράγματι, ε, το έργο μας επικεντρώνεται σε χώρες ε, όπου το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από κοινωνική και πολιτική αστάθεια. Και σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να ε, προχωρήσουμε σε ενδιάμεσες ε, μεσοπρόθεσμες πολιτικές. Όπως και να έχει όμως οι πολίτες θέλουν να δουν ποιο θα είναι το μέλλον τους, ιδίως στη χώρα προέλευσής τους. Παρά να πω ότι η μετανάστευση προκύπτει ακριβώς από αυτή την έλλειψη ελπίδας από στις χώρες προέλευσής τους. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και τη μετανάστευση υπό τη διάσταση των δεξιοτήτων Βεβαίω αναφέρομαι εδώ πέρα στην νόμιμη μετανάστευση. Χαίρομαι ιδιαίτερω που... Να αναφέρω ε, μια εκδήλωση που διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Επιτροπή για τους ε, ανέργους ε, στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπό τον έλεγχο και του συναδέλφου από την Γενική Διάθεση Άγκρη, ήταν η πρώτη φορά όπου υπήρξαν ε, τέτοιες ε, χώρες εταίροι, ε, με τη συμμετοχή βεβαίω και του ETF, που ανέλυαν την κατάσταση. Φανταστείτε ότι για πρώτη φορά το 2014 καταφέραμε σε κάποιες περιπτώσεις χωρών εταίρων. Για πρώτη φορά λοιπόν αναλύσαμε την κατάσταση, γιατί δεν είχαμε χρόνο να αναφερθούμε σε όσους δεν ανήκαν στον χώρο της εκπαίδευση και κατάρτισης. Γιατί η ανεργία είναι αυτή που ε, επικρατεί στις συζητήσεις. Και το πρώτο που θα θέλω να φέρω εδώ είναι η έλλειψη πληροφορίας. Οι χώρες ε, οργανώνουν τις πολιτικές τους ε, με ιδιαίτερα ασαφείς συνθήκε δεν έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε για να πάρουν τι αποφάσει του. Και αν ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι να διασφαλίσουμε ότι όλη η στήριξη για την ε, παραγωγή και συλλογή δεδομένων και την ε, διαμόρφωση πολιτική βάση των δεδομένων, evidence-based, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Ιδάλλω, οι αποφάσει αυτέ λαμβάνονται εντελώ αυθαίρετα και δεν αιτιολογούνται από στοιχεία. Δεύτερο θέμα εδώ. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το επίπεδο των ανέργων, των όσων δεν απασχολούνται, ε, στις χώρες όπου μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα, μόνο σε 11 από τις 13 ε, χώρες καταφέραμε να υπολογίσουμε αυτό τον αριθμό από στατική σκοπιάς δηλαδή σε όσους δεν συμμετείχαν στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, ο αριθμός λοιπόν είναι διπλάσιος από ό,τι στην Ευρώπη. Επομένω, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό απαιτείται άμεση ανάληψη δράσης για να μεριμνήσουμε, να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί που δεν ε, υπάγονται στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Γιατί πρέπει να περάσουμε πέρα από τα στατιστικά στοιχεία. Μιλάμε για ανθρώπους και να δούμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Έχει ήδη ξεκινήσει λοιπόν η συνεργασία με αυτές τις χώρες, θα συνεχίσουμε το 2014. Το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να περάσουμε από αυτή την ιδέα ε, της ε, αντιγραφή και επικόλυση λύσεων από τη μία χώρα στην άλλη ή να θεωρούμε ότι ένα μοντέλο θα ισχύει για όλου, πρέπει να έχουμε προσαρμοσμένε, ειδικά προσαρμοσμένε ε, λύσει και πολιτικέ. Όμω για να γίνει αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρξει και κοινωνική διάσταση σε οτιδήποτε κάνουμε. Δεν μπορούμε μόνο να επιμείνουμε στην οικονομική διάσταση. Σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση. Βεβαίω δεν μπορούμε να πούμε ότι στην οικονομική διάσταση έχουν επιτευχθεί όλα. αντιθέτω νομίζω ότι πρέπει να προτείνουμε να συνεχιστεί η ε, κοινή μας ε, περισυλλογή με τους εταίρους μας, ε, σε ποιους ε, κοινωνικούς τομείς κοινωνικής ανάπτυξης θέλουμε να επικεντρωθούμε, πού μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Γιατί δυστυχώς πρέπει να πω ότι υπάρχει οικονομική ανάπτυξη σε κάποιες χώρες, όπως η Τουρκία για παράδειγμα, αναφέρω και πάλι, όμως δεν μιλάμε ουσιαστικά για αύξηση των θέσεων εργασίας. Πρέπει λοιπόν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, αξιοπρεπούς απασχόλησης και να γίνονται σεβαστά και τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί δάλος μπορεί να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης της κατάρτισης, αλλά χωρίς όφελος. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να απάντησα ερωτήσεις. Κυρία Σχαντεχ. Ευχαριστώ. Ήταν ενδιαφέρον που άκουσα από εσάς ότι δεν αξιολογείται μονάχα τα επίσημα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αλλά και τα ανεπίσημα που είναι μια τεράστια θεά ζώνη στην ανάλυση των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των οργανισμών, αλλά βέβαια και στις εκλογικές περιφέρειες συχνά όταν τα λέω αυτά με ρωτούν μα πώς είναι δυνατόν να επαληθευτούν τα στοιχεία αυτά. Εγώ θεωρώ ότι ο οργανισμός σας εν προκειμένου έχει μεγάλη σημασία για την καλλιέργεια του εδάφους αυτού έτσι ώστε να προκύψουν κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες μέλη και τα όσα, απο... και τα όσα αποφασίζουμε εδώ να γίνουν απτά. Κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο και για την ισότητα των φύλων. Εάν σκεφτούμε δηλαδή πώς έχει η κατάσταση, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούμε και έχουμε γενναίες γυναικών, οι οποίες έχουν αποκτήσει δεξιότητες μέσω ανεπίσημης εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων τους μέσα από καταστάσεις που δεν αποτελούν επίσημη εκπαίδευση ούτε επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο έχουν, έχουν ε, αποκτήσει σημαντικές ικανότητες, σημαντικές δεξιότητες που δεν εμφανίζονται και δεν αναγνωρίζονται πουθενά. και όταν θέλουν να αναλάβουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό καθήκον αυτό να εκδώσετε συγκεκριμένες κατευθύνες γραμμές για το τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις ώστε να αναγνωρίσουν αυτές τις ε, γνώσεις. Εδώ θα με ενδιαφέρει να μάθω αν έχετε συγκεκριμένα σχέδια και ποια. Thank Σας ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σας που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ε, χώρες εταίρους όπως τονίσατε και εσείς. Γιατί δηλαδή είναι τόσο σημαντικό για τις χώρες εταίρους, διότι επιπροσθέτως των όσων συμβαίνουν σε ορισμένες χώρες μέλη, στις χώρες εταίρους, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουμε σημαντικό ανεπίσημο τομέα και εκπαίδευσης αλλά και της οικονομίας. Και όσοι και όσες βρίσκονται εκεί δεν έχουν προοπτικές σταδιοδρομίας διότι δεν υπάρχει αναγνώριση των επιτευμάτων τους. Έτσι λοιπόν μαζί με όλη τη δουλειά που κάνουμε σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, προσπαθούμε αμέσως να περιλάβουμε και άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί, για παράδειγμα την αναγνώριση της πρώτερης μάθησης στο ανεπίσημο πλαίσιο και όχι μόνο της ίδιας της μάθησης, που ίσως όπως είπατε και εσείς να μην είναι απαραίτητα μέσα στο επίσημο πλαίσιο, μπορεί να είναι και πάνω στη δουλειά. Υπάρχουν ναι, κατευθυντήρες γραμμές και καλές εμπειρίες στην Ευρώπη και εποφελούμεθα από αυτές. Υπάρχουν χώρες μέλη που είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους και να εξηγήσουν πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά. Ο μεγαλύτερος φόβος που έχουμε για την ώρα στις χώρες εταίρους είναι η έλλειψη οποιοδήποτε συστήματος εξασφάλισης της ποιότητας πιστοποίησης των δεξιοτήτων. Και γι' αυτό η δουλειά μας είναι σημαντική και για να διασφαλίσουμε ότι η ποιότητα θα μπορέσει και να εισαχθεί αλλά και να γίνει αντικείμενο διαχείριση στις χώρες εταίρους. Διότι υπάρχει κίνδυνος, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διαφθοράς, εκτός από ανθρώπους που πραγματικά είναι άξιοι και είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν τα προσόντα τους, να παράλληλα να έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα, έχουν, θα διαθέτουν κάποια πιστοποιητικά που δεν έχουν καμιά αξία. Δεν γνωρίζουν καν οι ίδιοι τι γράφει πάνω στα πιστοποιητικά. Γι' αυτό η δουλειά μας είναι τόσο σημαντική και είναι και διπλή η προσπάθεια. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι ούτε τιμωρούμε εκείνους που έχουν το δικαίωμα να αναγνωριστούν τελικά τα προσόντα τους, διότι η χώρα τους δεν έχει το απαραίτητο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, από την άλλη, από την άλλη πλευρά να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα συνεχίσουν να εκδίδονται πιστοποιητικά δεξιοτήτων όπως το παρελθόν. Οι πολίτες σε ένα βαθμό πληρώνουν και τις καταστάσεις του παρελθόντος. Παράδειγμα αραβικών χωρών, όπου οι στόχοι της χιλιετίας ζητούσαν από τις χώρες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στην στοιχειώδη εκπαίδευση. Και πρόσβαση μάλιστα αν είναι δυνατόν και μετά από την στοιχειώδη εκπαίδευση, από την ποσοτική άποψη όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν και οι στόχοι εκπληρούνται και όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Όμω δυστυχώ η ποιότητα των επιτεύξεων αυτών είναι τόσο χαμηλή και οι άνθρωποι δεν αποκτούν προϊόντα, ε, δεν αποκτούν προσόντα και δεξιότητε στην επαγγελματική εκπαίδευση, δεν έχουν τη βάση. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να επεκταθεί αυτή η πρακτική έκδοση πιστοποιητικών και διπλωμάτων που δεν καλύπτουν πραγματικά προσόντα με νέο σημείο εισόδου που θα είναι έκδοση πιστοποιητικών για την ανεπίσημη εκπαίδευση. Να μην ανοίξουμε και άλλο παράθυρο δηλαδή. Δεν υποτιμώ καθόλου αυτό που λέτε πάντως, ιδιαίτερα εκείνες και εκείνοι που δεν είχαν, εκπαίδευση, ε, πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση, όπως έχουμε και στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης όπου δεν είναι μόνο οι νέοι, αλλά και οι πολύ νεαροί δηλαδή, αλλά και οι ενήλικοι, έχουν πολλοί από αυτούς αποκτήσει πολλές γνώσεις και δεξιότητες, δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να τις πιστοποιήσουν. Γι' αυτό εργαζόμεθα από αυτού. Δίνουμε προτεραιότητα ιδίως στις χώρες εκείνες οι οποίες διαθέτουν ήδη συμφωνίες Mobility Partnership υπογραμμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνουν επομένως στην ε, νόμιμη μετανάστευση και θέλουμε εκεί να υπάρξει μια αξιοπρεπής αναγνώριση των δεξιοτήτων τους εφόσον αποφασίσουν να βγουν στο εξωτερικό και να εργαστούν εκεί. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν το θέμα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του ETF. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Επιθυμεί άλλος κανείς. Δεν βλέπω άλλα χέρια. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, αγαπητή κυρία Σερμπάν, κυρία υποψήφια. Σας ευχαριστώ. Δεν μας μένει καμιά αμφιβολία για τον δίκαιο χαρακτήρα της ε, πρότασης που γίνεται από το Συμβούλιο Διοικητών της ε, οργάνωσης. Ως Κοινοβούλιο έχουμε δει και την προσωπική σας δέσμευση και την ποιότητα των αναλύσεών σας, την ικανότητα να συγκεντρώσετε έναν αριθμό φορέων ε, γύρω σας και την στήριξη του Κοινοβουλίου. Και όταν μιλώ για εδώ, εννοώ το Κοινοβούλιο, βλέπουμε εδώ λοιπόν τον ρόλο των οργανισμών καμιά φορά να αμφισβητείτε ε, καμιά φορά και από την άποψη της αρχής των, της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό. Σεις όμως καταδεικνύεται ποιο μπορεί να είναι και το θετικό έργο ενός οργανισμού και μάλιστα σε περίοδο όπου τα γεγονότα σε αυτό που αποκαλούμε κάπως αυθαίρετα γειτονικέ χώρες ενισχύουν, επιβεώνουν την ποιότητα της εντολής σας. Όλοι θα θυμάστε ότι έχετε κληρονομήσει την συνομοσπονδία που είχε ονειρευτεί ο Φρανσουά Μιτεράν με την ιδέα ότι στο περιθώριο της Ευρώπης θα δημιουργούνταν ένας χώρος όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δημιουργήσει συνεργασίες de facto με μια πραγματική καθημερινή διπλωματία. Και όταν μιλήσατε άκουσα κάτω από τα όσα λέγατε αυτή την πραγματικότητα να εξακολουθεί να είναι ζωντανή. Σε μια περίοδο όπου βλέπει κανείς ότι η κλασική ας πούμε διπλωματία αν και στο επίπεδο της Ένωσης δεν υπάρχει κλασική διπλωματία αλλά τέλος πάντων η διπλωματία στις κλασικές της εκφάνσεις αντιμετωπίζει σκληρά εμπόδια. Ό,τι λοιπόν μπορεί να κάνει ο οργανισμός σας δεν μπορεί παρά να ευνοήσει αυτή τη συνειδητοποίηση και αυτή την ε, ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος στην στρατηγική προσέγγιση αυτών των γειτονικών χωρών που εμπίπτουν τις αρμοδιότητες του οργανισμού σας. Από όλα λοιπόν τα μέλη μας σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω το λόγο βεβαίω για να ολοκληρώσετε εσείς την συζήτηση αυτή και θα πω και δύο λόγια για την διαδικασία μετά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Τι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ και όχι μοναχά για την σημερινή ημέρα, αλλά και για τα πέντε χρόνια, πέντε χρόνια εντατικής εργασίας. Λέμε στον οργανισμό μας ότι κάνουμε πραγματικά αυτό που αγαπάμε και βλέπουμε την χρησιμότητα του οργανισμού μας. Και είμαι βέβαια ότι και εμείς και εσείς αλλά και έξω από την αίθουσα αυτή πολλοί βλέπουν τον TTF ε, σαν οργανισμό που είναι πολύ χρήσιμος. Φτάνουμε στην 20 ετία του οργανισμού μας, στην 20 ετία επέτειο που μας θυμίζει, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, το 89, 89 και αρχές του 90, όταν λήφθηκε η απόφαση για τη δημιουργία του οργανισμού μας, ως συνέπεια των αλλαγών των γεωγραφικών συνόρων της Ένωσης, με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί ανάμεσα στις χώρες μέλη και σε έναν πολυπολικό κόσμο ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο πώς θα συνεργαστούμε. Ωστόσο φέτος 2014, 2014 είναι και η εκατοστή επέτειος όπου σε, ένα από, σε μια από τις χώρες εταίρους της ETF, δηλαδή το Σαράγεβο, ξεκίνησε εκείνος ο τρόμερος πόλεμος. Βεβαίως και σε άλλες χώρες τέρους ε, δεν υπάρχει μεγάλη σταθερότητα. Χρειαζόμαστε ωστόσο την ειρήνη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χέρι με χέρι. Ένας λόγος που έχω τέτοια εμπιστοσύνη στο έργο ολοκλήρωσης της Ένωσης είναι ότι θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε αυτή τη συνεργασία και με τις γειτονικές μας χώρες. Και ο οργανισμός μας θα είναι εκεί για να εξασφαλίσει την πορεία αυτή είτε με εμένα ως διευθύντρια είτε και χωρίς εμένα. Πάντως εγώ είμαι απόλυτα ε, δεσμευμένη να συνεχίσω το έργο μου. Ευχαριστώ. Το γνωρίζουμε λέει η Πρόεδρος. Και σας, ευχαριστούμε πολύ για τη συνέχεια της διαδικασίας. Να σας πω ότι θα γράψω μια επιστολή στο Σύμβουλο των Δικητών για τον ενημερώσω για την ακροασή σας και να πούμε και την άποψή μας για την πρότασή τους. Η επιστολή σαφώς και θα διανεμηθεί στους συντονιστές για να συνεισφέρουν και αυτοί αν το επιθυμούν ή να διορθώσουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι διάδοχοί μας εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης θα έχουν την ευκαιρία να έχουν μια καρποφόρα συνεργασία μαζί σας και σας εύχομαι εκ μέρους και όλων των συναδέλφων μια πολύ καλή νέα θητεία και αν ε, μείνετε για την επόμενη μισή ώρα, σας καλώ ε, να μείνετε εδώ για το τελευταίο ποτό που θα πιούμε, γιατί είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο Παρουσίασε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις πρότασεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης ε, Ιανουαρίου. Πρόκειται για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης, πρόσβαση των εργαζομένων στις υπηρεσίες κινητικότητας και συνέχιση της ολοκλήρωσης των αγορών εργασίας. Η πρόταση αυτή για το Γιούρες είναι τμήμα ε, μια σειρά μέτρων που λαμβάνονται για να ε, βοηθήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των όσων συζητήσαμε προηγουμένως ε, και για τα οποία έχουμε ακόμα μια δυσκολία με την ελληνική προεδρία και μια διάταξη την οποία εγκρίναμε στη διάρκεια της διαδικασίας προπολογισμού στην έκθεση EASY. Ε, στους συντονιστές αποφασίσαμε να μην υπάρχει εισηγητής για το θέμα αυτό, διότι ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεδομένου ότι παρουσιάστηκε με μεγάλη καθυστέρηση η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι την πρόταση αυτή την αναμέναμε εδώ και αρκετό καιρό και ε, κάποιες πρωτοβουλίες, κυρίως η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ε, είχε αν γίνει με την προοπτική της παρουσίασης ε, αυτής της πρότασης και έτσι οι συντονιστές αποφάσισαν να αφήσουν ε, ε κενό το θέμα αυτό και να το παραδώσουν στους διαδόχους μας αλλά από την άλλη θεωρήσαμε ότι είναι κρίμα να μην παρουσιάσει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επομένως θα έπρεπε να της δώσουμε τη δυνατότητα να ενημερώσει την Επιτροπή του Κοινοβουλίου για το περιεχόμενο αυτής της πρότασης και ε, τη σημασία που ε, έχει και που θα έπρεπε να μας οδηγήσει. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κιμωρά, ο οποίος είναι τμήματάρχης του Τμήματος Απασχόλησης και Κινητικότητας, για να μας παρουσιάσει την πρόταση κανονισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την παρουσίαση της πρώτης της Επιτροπής για το EURES. Θα ήθελα συντομία να σας παρουσιάσω κάποια ε, στοιχεία ε, για την πρόταση αυτή και μετά να σας πω πέραν του ευρύτερου πλαισίου και τις γενικές γραμμές προσανατολισμού. Το ευρύτερο πλαίσιο βασιζόμαστε στο άρθρο 46 της συνθήκης που ε, παρέχει αρμοδιότητες, εξουσιοδότηση για τη θέσπιση μηχανισμού που φέρνει σε επαφή τον τομέα της προσφοράς και της ζήτησης και αυτό συνδέεται με το άρθρο 45 που προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να μετακινούνται και να ζουν και να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις βάση της εθνικότητάς τους. 492 του 2011 είναι ε, η βάση μας αυτός ο κανονισμός ε, που συνδέεται και μια πρόταση οδηγίας που έγινε ε, ε, προσφάτως ε, για την εφαρμογή και την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Το Euros ισχύει εδώ και μερικά χρόνια. Θεσπίστηκε για να επιτρέπει στους εργαζόμενους ενός κράτους μέλους ε, να λαμβάνει πληροφορίες για την διάθεση, την προσφορά θέσεων απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος και αντιστοίχως να επιτρέπει σε εργοδότες ενός κράτους μέλους να έχει πρόσβαση στα βιογραφικά σημειώματα ετούντων απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος. Συνδέεται με τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, επιτρέπει ε, χάρη σε αυτή την ε, Ιντερνετική πύλη να ξεπερνώνται τα γλωσσικά και άλλα εμπόδια. Σήμερα έχουμε περίπου 2 ε, με 3 εκατομμύρια αποτελέσματα, δηλαδή επισκέψεις σε αυτή την πύλη κάθε μήνα. Και υπάρχουν χιλιάδες ε, ε, μέλη της ε, πύλης που επιτρέπουν αυτή την σύνδεση προσφοράς και ζήτησης. Έχει, διαθέτουμε και ένα δίκτυο 900 συμβούλων που επιτρέπουν αυτή την επαφή, την δημιουργία επαφής και τελικά σε χιλιάδες προσλήψεις. φαίνεται ότι παρά την ε, επιτυχία αυτής της πύλης ε, δεν αξιοποιείται παρκώς. Πρόκειται πάντα βεβαίως για αποφάσεις μεμονωμένων ατόμων που πρέπει να επιλέξουν ε, να αξιοποιήσουν αυτό το μέσο. Βλέπουμε όμως ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο μεγάλων οικονομικών αποκλήσεων, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, στον, ε, στο ποσοστό ανεργίας, ε, που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 27% από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, βλέπουμε ότι αντιστοίχω διαμορφώνεται και το τοπίο σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των εργαζομένων. Για να σα δώσω και ένα στοιχείο, όταν ρωτάμε του Ευρωπαίου πολίτε ε, ποιε είναι οι προθέσει του ό,τι αφορά την κινητικότητα, το 20% απαντά ότι του ενδιαφέρει η διασυνοριακή αυτή κινητικότητα. Σε αυτό το 20% ένα σημαντικό τμήμα, 1,2% των πολιτών δηλαδή, μας λέει ότι έχω πραγματικά την πρόθεση να μετακινηθώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Έχουμε λοιπόν ε, ένα λόγο 1 προς 5 για τα άτομα που θέλουν να μετακινηθούν μέσα στη χρονιά. Και έχουμε αντίστοιχο ε, ζήτημα με τους ε, εργοδότες. Βλέπουμε ότι το 40% των ε, εργοδοτών λένε ότι έχουν, αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν εργαζομένους που έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και βεβαίως και με την δημογραφική αλλαγή σημαίνει ε, μείωση κατά 18.000 ε, εργαζομένων μέσα στα επόμενα 20 έτη. Επομένως θα υπάρχει αυτή η έλλειψη εργατικού δυναμικού που θα γίνεται όλα ένα και πιο εμφανής. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις διαπιστώσεις και παρά την ε, ελκυστικότητα αυτού του μηχανισμού φαίνεται ότι πρέπει να ενισχύσουμε το EURES για να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί περαιτέρω και να βοηθήσει για την ενίσχυση της ε, ενιαίας αγοράς εργασίας. Η πρόταση της Επιτροπής λοιπόν έχει ως στόχο την, να επιτρέψει αυτή την ενίσχυση και ε, να συγκεκριμενοποιήσει ε, την νομική βάση του Γιούρες βάσει του κανονισμού 492 του 11 και της ε, απόφασης τη Επιτροπής της 16 η ε, Νοεμβρίου 2012. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ε, πρότασης, θα ήθελα να επισημάνω τα εξή στοιχεία. Πρώτο, σημείο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόλου του Γιούρες έχει ως στόχο να προσαρμοστεί καλύτερα ε, το Γιούρες στην ε, ε, λειτουργία της αγοράς, να ενσωματωθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις οι δυνατότητε επικοινωνία και ανταλλαγή ε, δεδομένων, να ε, λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι υπάρχουν ε, εξελίξει στην αγορά εργασία και έτσι στα άρθρα 14-17 προβλέπουμε την θέσπιση μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και έτσι να ενισχύσει τη διαδραστικότητα με τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, μεταρρύθμισης είναι να επιτρέψουμε να προβλέψουμε το Γιούρες να έχει μια πιο ολοκληρωμένη ανταλλαγή και διευκόλυνση των επαφών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, ε, κοινοποιούν όλες τις ε, προσφορές θέσεις εργασίας ε, στο Γιούρες. Και έτσι υπάρχει και αυτός ο περιορισμός στη δυνατότητα πρόσβαση στην πληροφορία. Σε ό,τι αφορά τις ε, θέσεις απασχόλησης που μένουν κενές και θα μπορούσαν να πληρωθούν από κάτι άλλου κράτους μέλους. Αυτές οι διοικητικές, διοικητικοί περιορισμοί θα πρέπει να αρθούν στο πλαίσιο της πρώτας κανονισμού. Είναι όλα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 14 της πρότασης. η αύξηση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης συνδέεται και με την ενίσχυση της ε, δυνατότητας ε, αντιστήχησης ε, των, της προσφοράς και της ζήτησης απασχόλησης. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και μια προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί στον τομέα της ταξινόμησης. Όλα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 16 της πρότασης όπου πρέπει να υπάρχει μία αυτόματη αντιστοίχηση μεταξύ της προσφοράς αφενός και της ζήτησης, δηλαδή των ε, βιογραφικών σημειωμάτων. Όλα αυτά βασίζονται στο ΕΣΚΟ και θα μας επιτρέπουν να περιγράψουμε και τη θέση απασχόλησης που παρέχεται αλλά και τις ε, δεξιότητες που απαιτούνται και ποιε είναι από την άλλη μεριά και οι δεξιότητε που κρύβονται πίσω από τα βιογραφικά σημειώματα. Να υπάρχει λοιπόν μια καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ των δύο αυτών πηγών πληροφόρηση. Τέταρτο στοιχείο ενίσχυση, που προβλέπεται στα άρθρα 18-24 της πρότασης κανονισμού αφορά την ε, ανάπτυξη υπηρεσιών. Αυτή η έννοια των υπηρεσιών και για τους, ε, αυτούς που ψάχνουν μια θέση απασχόληση και για τους ε, εργοδότες είναι κάτι νέο, ένα νέο στοιχείο δεν υπήρχε προηγουμένως. Θέλουμε να ευνοήσουμε ε, αυτή την κινητικότητα με όλα τα παραλυκόμενα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, την ενημέρωση όσων ζητούν μια θέση εργασίας ή και από την πλευρά των εργοδοτών άλλη πτυχή αφορά τις εταιρικές σχέσεις και τη διεύρυνση του δικτύου Γιούρες πέραν των ε, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης μέσω διαδικασιών που αναφέρονται στο κανονισμό με ποιοτικά κριτήρια που επιτρέπει τη διεύρυνση ε, των εταιρικών σχέσεων και με ιδιωτικούς φορείς ή με άλλους εταίρους που ε, προσδιορίζονται σε εθνικό πλαίσιο. Σήμερα ε, αυτές οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ε, μεταφέρουν περίπου το 30% του όγκου δεδομένων για την ε, προσφορά και ζήτηση απασχόλησης. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει και μέσω περαιτέρω εταίρων. Στα άρθρα 3 13 του κανονισμού ε, προβλέπονται αυτά τα ζητήματα εταιρικών σχέσεων. Τελευταίο σημείο ο νέος κανονισμός εισάγει σαφείς ε, κανόνες που επιτρέπουν στην Επιτροπή να ασκεί εξουσίες, ε, εκτελεστικές εξουσίες, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον μορφότυπο των πληροφοριών που επιχάνουν ανταλλαγή μεταξύ των υπηρεσιών, αλλά και ε, αρμοδιότητες επικαιροποίησης των εταίρων γιούρες. Στο άρθρο 33 του κανονισμού προβλέπονται όλα αυτά. Αυτά εν ολίγης, ήθελα να σας πω. Στόχος μας εδώ είναι να έχουμε ένα νέο εξυγχρονισμένο μέσο στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων για καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Αυτή η πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να αντικαταστήσει το, άρθρο, το κεφάλαιο 2 του 492-2011 καθώς και το άρθρο 38 του ίδιου κανονισμού ε, ε, εκεί πέρα δεν υπήρχε κοινή αντίληψη μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και αντικαθιστά και το 233 και τον ε, χάρτη του Γιούρες. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι συνθέτουμε όλες αυτές τις διαφορετικές υφιστάμενες πηγές. Διαμορφώνουμε μια νέα ενιαία βάση και προτείνουμε και κάποια σημεία βελτίωσης που μόλις σας ανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Διαβάσατε τη σκέψη μου γιατί είχα δει ότι ε, υπάρχουν 37 άρθρα στο σχέδιο κανονισμού και σκεφτόμουν ότι πρέπει να ευχηθώ καλή τύχη σε όσους αναλάβουν την διαπραγμάτευση του κειμένου, γιατί παρότι μιλάτε για σύνθεση και εξορθολογισμό ε, στοιχείων που υπάρχουν ήδη, ε, δεν αλλάζει το γεγονό ότι πρόκειται για ιδιαίτερα μακροσκελέ κείμενο. Και επομένω ε, θα είναι δύσκολη η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Λουβιεύσκα, παρακαλώ. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εξετάζοντα το Γιούρες, ορισμένε φορέ όταν έμπαινα στην ε, δικτυακή πύλη είχα την εντύπωση ο λειτουργεί ότι λειτουργεί με βάση γλωσσικές δεξιότητες. Γνωρίζουμε ξένες γλώσσες, είτε ενεργητική είτε παθητική γνώση των γλωσσών, είτε έχουμε παθητική γνώση, τις οποίες γνωρίζουμε και δεν τις χρησιμοποιούμε, ή ενεργητική γνώση και χρήση της γλώσσας αλλά εδώ ε, φαίνεται ότι λειτουργούν τα πράγματα ως παθητική γνώση της γλώσσας. Λέτε ότι λαμβάνετε προφορές από τα κράτη-μέλη, λέτε ότι θα πρέπει να έχετε περισσότερες θέσεις εργασίας, να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας, αλλά κατά την άποψή μου, προκειμένου να μπορέσετε να αντιστοιχίσετε τις ανάγκες της ε, αγοράς εργασίας με τις ανάγκες των εργοδοτών, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο. Και πολύ φοβάμαι ότι οι προτάσεις σας δεν θα πληρώσουν το κενό που υπάρχει. Δεν θα ανταποκριθούν στους όρους των, εργαζομε... των εργοδοτών που συγγνώμη, των εργαζομένων που ενδιαφέρονται για τις προσφορές, να κατανοήσουν ποια είναι η προσφορά της θέσης εργασίας και φυσικά οι εργοδότες δεν θα μπορούν να αντιληφθούν ποιους εργαζόμενους χρειάζονται στο μέλλον. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Αυτό που προτείνεται προβλέπεται να ε, περιλαμβάνει και κάποιες ε, ε, εταιρικές σχέσεις με εργοδότες που θα χρησιμοποιούν συστηματικά το σύστημα και θα ενημερώνουν τακτικά για θέσεις εργασίας, για νέες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν ή θα σταματήσουν να προσφέρονται σε μια επιχείρηση θα υπάρχει κάποιος ο οποίος ε, θα σας συμβουλεύει, θα συμβουλεύει το σύστημα και θα συμβουλεύει και τους εργαζομένους εάν ε, αν ενδιαφέρονται για μια θέση εργασίας. Λέτε ότι ένα 20% ενδιαφέρεται για κινητικότητα, αλλά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 0,2% λέτε μετακομίζει σε μια άλλη χώρα. Γιατί λοιπόν υπάρχει ένα 20% το οποίο θέλει να αλλάξει χώρα και τελικώς ε, δεν μεταφέρεται. Θα πάρουμε όλες τις ερωτήσεις μαζί και θα απαντήσετε συνολικά. Η Γιούτα Στάνχομ και μετά η κυρία Σουρέτερ. Ε, ευχαριστώ. Πρώτα να σας ευχαριστήσω για τις εξηγήσεις που δώσατε. Είμαι βεβαία ότι η πρότασή σας θα προσφέρει πολύ ε, τροφή για συζήτηση και στην επόμενη δύο κοινοβουλευτική περίοδο. Σημαντικό βρίσκω να ξεκαθαρίσουμε ότι μόνο με την κινητικότητα των εργαζομένων δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα της μεγάλης ανεργίας στην Ευρώπη. Εσείς θέλετε να βελτιώσετε την κινητικότητα των εργαζομένων για να καταπολεμήσετε την ανεργία. Αυτό για μένα δεν θα είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό. Μιλήσατε επίσης, αν κατάλαβα καλά, για την επιθυμία σας ε, με την πλατφόρμα να φτάσετε σε 2.500 διαμεσολαβήσεις το χρόνο. Ο αριθμός αυτός μου φαίνεται πάρα πολύ μικρός εν ώψη της μεγάλης προσπάθειας που προηγείται. Από την δική μου σκοπιά η πρότασή σας αγνοεί τα μεγαλύτερα εμπόδια για την κινητικότητα και ιδίως για την διαμεθοριακή κινητικότητα και οι αριθμοί που αναφέρατε σε αυτούς μάλλον βρήκα να λείπει και πόσες εργαζόμενες και εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται διαμεθοριακά μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή κατοικούν σε μια χώρα, εργάζονται σε μια άλλη. Εκτός από τις γλωσσικές γνώσεις εκεί βέβαια και την έλλειψή τους, ένα ρόλο παίζει και η έλλειψη ενημέρωση για την εργασιακή νομοθεσία, κοινωνική νομοθεσία και ούτω καθεξής, που είναι απαραίτητο να είναι γνωστή. Γιατί αυτά θεσπίζονται διμερώς από τις δύο χώρες. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διακινούνται διαμεθοριακά έχουν και τα μεγαλύτερα εμπόδια. Και μάλλον τελικά υφίστανται μειονεκτήματα παρά να εποφελούνται από τα πλεονεκτήματα και όταν η ενημέρωση γίνεται ακόμα χειρότερη δεν ωφέλει σε τίποτα η προσπάθεια διαμεσολάβησης. Για μένα η παροχή συμβουλών και η ενημέρωση είναι κεντρικά θέματα για να εξελιχθεί η κινητικότητα των εργαζόμενων. Εμείς θέλουμε όμως δίκαια και έντιμη διαμεθοριακή απασχόληση, όχι εκμετάλλευση. Εάν στο μέλλον η προσπάθειά σας περιοριστεί μονάχα στη διαμεσολάβηση, έχω ορισμένες ερωτήσεις. Δηλαδή, τι λέτε για την στάθμιση της ποιότητας των χωρών μελών, ε, για τις ποιότητες συγγνώμη, των θέσεων εργασίας και τον ρόλο των ε, συμφωνιών μεταξύ κοινωνικών εταίρων, αλλά και αυτών που διαμεσολαβούν στην ε, παροχή υπηρεσιών, που μέχρι τώρα στην πρόταση σας περιλαμβάνονται μονάχα προαιρετικά. Εξάλλου, η ΕΟΡΕΣ μπορεί να παίξει και ένα ρόλο για την εκπλήρωση της ε, εγγύηση για τους νέους, για την νεολαία δηλαδή, της απόφασης δηλαδή του Συμβουλίου του 2012 για τις ε, πρακτικές ασκήσεις. Πρακτική άσκηση όμως χωρίς θέσεις εργασίας που να συνοδεύονται από κοινωνικές διασφαλίσεις. Απλώς δηλαδή θα πρόκειται για ε, νεαρούς εργαζόμενους οι οποίοι διακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη για να προσφέρουν εργασία υπό ε, μειονεκτικές συνθήκες για την εγγύηση για την νεολαία επίση μα ενδιαφέρει η απασχόληση αυτή να είναι ποιοτικά υψηλή ποιότητα. Έχω και τρία ακόμα ερωτήματα. Θέλω να μάθω εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την συμπερίληψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στον κανονισμό, όπως, τον έχουμε, όπως την έχουμε και στον γενικό κανονισμό, και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και η δεύτερη ερώτηση προβλέπεται η διαμεθοριακή διακίνηση και στον κανονισμό ότι ωραίες. Και τέλος οι αρμοδιότητες για την υποβολή αιτήσεων, για την διαχείριση των κοντιλίων και για τον συντονισμό θα παραμείνουν αυτά ως αρμοδιότητες των περιφερειακών αρχών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε ακόμα δύο εγγεγραμμένους και μετά θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Πρώτον, η κυρία Σρέντερ. Οι ερωτήσεις μου ακολουθούν αυτές τις ε, προαλυσάσεις, διότι πραγματικά βλέπω να λείπει αυτές οι εταιρικέ σχέσεις, οι partnerships δηλαδή, που είναι η καλύτερη δυνατότητα για την διασφάλιση απασχόλησης, φαίνεται στον νέο κανονισμό να μην παίζουν ρόλο. Και αυτό με δυσαρεστεί πολύ, το λέω ειλικρινά, διότι ένα, ευρωπαϊκό, ένα κεντρικό ευρωπαϊκό στοιχείο επιτόπου έφνης αγνοείται. Η κινητικότητα, για παράδειγμα από το Παρίσι στο Βερολίνο, θα είναι σίγουρα πολύ μικρότερη ανάμεσα σε δύο μικρές ε, πόλεις εκατέρωθεν των πολωνογερμανικών συνόρων. Για κάντε μια σύγκριση των αριθμών και θα δείτε τότε τα, γερμαν, τα γερμανοπολωνικά σύνορα άλλωστε δεν είναι και τα σύνορα που διέρχονται οι περισσότεροι. Για παράδειγμα τα γάλλο-γερμανικά σύνορα τα διέρχονται πολύ περισσότεροι για να εργαστούν. Και αυτά φαίνεται για εσά να μην παίζουν κανένα ρόλο. Θα δείτε άμα τα μελετήσετε αυτά τι μεγάλε διαφορέ υπάρχουν. Και εδώ τα πράγματα είναι πολύ στραβά μέσα στον κανονισμό που δεν απηχεί καθόλου τις πραγματικότητες στην Ευρώπη. Εδώ μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια ε, πολωνική πόλη και θέλουν να πάνε να εργαστούν στην Φραγκφούρτη ή και κοντά στην, ε, στα σύνορα όπου το βράδυ μπορούν να επιστρέψουν στις εστίες τους. Για πηγαίνετε λιγάκι στην ε, Φραγκφούρτη, στον Όντερ, όταν έρχονται τα τρένα και ακούστε λίγο πόσες γλώσσες μιλούνται εκεί και θα καταλάβετε τότε ποια είναι η πραγματικότητα της κινητικότητας στην Ευρώπη. Και αυτά που σκέφτεστε εσείς εδώ ότι μπορεί κάπου μακριά ή με ένα, με ένα ε, ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορείτε να βοηθήσετε οι άνθρωποι να πάνε από το Παρίσι στο Βερολίνο ή από το Βερολίνο στην ε, Βαρσοβία, αυτά είναι πράγματα της φαντασίας. Αν δω και την Ουγγαρία μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας ή και Σλοβακίας, εκεί οι διακινήσεις είναι πολύ εντονότερες, διότι βεβαίως και η γλωσσική φραγμή είναι πολύ χαμηλότερη. Εκεί είναι οι πραγματικότητες όπου πρέπει να μπει μέσα η διαμεσολάβηση. Εκεί χρειάζεται ο Εύρες τα άλλα, αυτά που λέτε εσείς, είναι πολύ μικρό ποσοστό και εσείς τα κάνετε ακριβώς ανάποδα. Οι άνθρωποι επιτόπου δεν σας καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που θέλω να σας πω. Και το δεύτερο είναι ένα κεντρικό στοιχείο. Και πάλι επανέρχομαι σε αυτά που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Ένα κέριο στοιχείο της διαμεσολάβησης αυτής σήμερα εν ώψη του γεγονότος ότι γίνεται τόσο μεγάλη πίεση μέσω της διαμεθοριακής διακίνησης στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Οι άνθρωποι στην διαμεσολάβηση που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να είναι βέβαιοι ότι πάλι εκεί δεν πρόκειται να τους εξαπατήσουν και να ε, τα δικαιώματά τους. Και όχι μόνο για το ευαίσθητο θέμα της απόσπασης, ή για το ακόμα πιο ευαίσθητο θέμα των πρακτικών ασκήσεων. Τα εξετάζετε αυτά εσείς ως ε, ποιότητα. Μιλώ και για τα πολύ κλασικά ερωτήματα. του 2004-883. Αυτή η διαμεσολάβηση που κάνετε εσείς πηγαίνει παράλληλα και με μία ενημέρωση του προσωπικού όπου οι ερωτήσεις που θα σας κάνουν θα είναι ακριβώς αυτές και όπως εσείς θα μπορείτε να απαντήσετε. Αυτό είναι το συν του ΕΟΡΕΣ, όχι το ίντερνετ. Δεν χρειάζεται ολόκληρος οργανισμός ΕΟΡΕΣ για να ψάξω στο ίντερνετ να βρω ποια επιχείρηση μπορεί να χρειάζεται τι δεξιότητέ μου στην Γερμανία, στην Πολωνία, στη Γαλλία. Δεν χρειάζεται ο Η προστιθέμενη αξία του έωρε είναι να ξεκαθαρίσει τον κόσμο ποια κοινωνικά δικαιώματα έχει και πώς μπορεί να τα διασφαλίσει. Αν δεν τα κάνετε αυτά, τότε ολόκληρο το δίκτυο δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Έχοντας κατά νου τις ε, κοινέ μας προσπάθειε ε, πρόσφατα σε άλλη οδηγία. με λιγάκι, πρέπει να πω. Κοιτάζοντα το άρθρο 20, 22, 23, ακόμα και το άρθρο 7. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει αλληλεπικάλυψη εδώ μεταξύ του κανονισμού και της οδηγίας. Επομένω έχω την εξής απλή ερώτηση. Ε, θα υπάρξει συγχώνευση αυτών των υπηρεσιών, γιατί οι, οι υπηρεσίες στήριξης για τους εργαζομένους είναι για να παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και ούτω καθεξής. Ακριβώς ε, το ίδιο σχεδόν με αυτό που έχουμε πει στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Θυμάμαι και την ε, σφοδρή μας αντιπαράθεση για τα εθνικά σημεία επαφής και τον εθνικό συντονισμό. Και χαίρομαι ιδιαίτερος που αυτή τη φορά μιλάτε για εθνικά γραφεία συντονισμού. Όμως ε, και πάλι έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε αυτά τα δύο. Βεβαίως, γνωρίζω ότι αυτά τα εθνικά γραφεία συντονισμού έχουν και άλλες αρμοδιότητες και άλλα καθήκοντα πέραν των όσων ε, αναγράφονται στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία. Όμως, υπάρξει, υπάρχει σαφής αλληλεπικάλυψη. Επομένως, ε, εσείς τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Alors, ε, Λοιπόν, να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Έχει ήδη ξεκινήσει λοιπόν ο διάλογος και επί της ουσίας. Εγώ θα ήθελα μόνο να θέσω ένα πιο τοπικό ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει να εργάζεται επί του Γιούρες σε μια βάση την οποία εμείς αμφισβητήσαμε και μάλιστα φτάσαμε μέχρι και το δικαστήριο. Η Επιτροπή όταν υπέβαλε αυτή την πρόταση ήθελε ε, το Κοινοβούλιο να αποσύρει την πρότασή του. Ε, που αγνοούσε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Ποια είναι η γνώμη σας από αυτού, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από μια καλή βάση. Και οι διαπραγματεύσεις για αυτόν τον κανονισμό να μην χρειάζεται να περάσει μέσα από δικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφεραν για οι συνάδελφοι, αλλά ίσως και εσείς αν έχετε μια προσωπική γνώμη θα ήταν ε, χρήσιμο και για μας και για τους διαδόχους μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. La première question sur... Euh, Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, το γεγονός δηλαδή ότι το Euros δεν θα πρέπει να είναι πολύ παθητικό στις απαντήσεις του, αλλά πιο δραστήριο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην πρόταση, τα οποία στόχο έχουν ακριβώς να ενισχύσουν τη δυνατότητα ε, δράσης και μάλιστα προληπτικά, κυρίως σε θέματα τα οποία σχετίζονται με παροχή πληροφοριών, Ε, στοιχεία τα οποία εισάγουν μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες ε, θα προσφέρονται και στους εργοδότες αλλά και όσους αναζητούν θέση εργασίας. Να μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο και με περισσότερες λεπτομέρειες πριν, στη διάρκεια και μετά ε, της διαδικασία κινητικότητας και ε, η έννοια αυτής της εταιρικής σχέσης που αναφέρατε στα όσα μας είπατε, τα οποία θα πρέπει ε, να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Γιούρες και ε, φυσικά ε, εάν πρόκειται και διαμεσολάβηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θα μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο μετά την θέση εφαρμογή του κανονισμού. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να δραστηριοποιηθεί περισσότερο το Γιούρε και περιλαμβάνονται εδώ στην πρόταση. Όσον αφορά το θέμα των εμποδίων, όντως ε, υπάρχουν αρκετά εμπόδια τα οποία ε, μας ενδιαφέρουν κυρίως στην διασυνοριακή κινητικότητα. Υπάρχει κυρίως το πρόσκομα της γλώσσας. Ε, εξετάζουμε και τα αποτελέσματα του ευρωβαρομέτρου και αυτό είναι στην πρώτη θέση. Αλλά αμέσω μετά ακολουθεί το γεγονός ότι ε, κάποιος μπορεί να μην βρει μια θέση εργασίας. Ξέρουμε ότι το βασικό κίνητρο για να αλλάξει κάποιος χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια θέση εργασίας. Πρόκειται για το κύριο κίνητρο της κινητικότητας. Και αυτό το πρόσκομα εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό σήμερα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά κίνητρα για την κινητικότητα και σας ανέφερα και τα, η διαφορά των ποσοστών απασχόλησης και το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχει προσφορά η οποία δεν καλύπτεται από τη ζήτηση. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε και αυτή τη διάσταση ε, και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόσκομα ε, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για να αποκτήσει κάποιος μια θέση εργασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος και το ε, EURES είναι ένα εργαλείο σε αυτή την περίπτωση το οποίο μας βοηθά να δίνονται σε διεθνές επίπεδο στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή δίνονται σε εθνικό επίπεδο. Ε, δημοσιοποιούνται οι θέσει εργασία σε εθνικό επίπεδο, αλλά η ιδέα είναι να υπάρχει και κάλυψη ε, πέραν των, ε, του 30% των θέσεων εργασίας που δίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα. όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων που αλλάζουν χώρα, καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Υπάρχει ο κανονισμός ο οποίος καλύπτει επαρκώς το γεγονός ότι ο εργαζόμενος ο οποίος θα μεταμαναστεύσει βάσει της συνθήκης έχει τα ίδια δικαιώματα και την ίση, δικαίωμα ίσης μεταχείρισης. Και ε, ο κανονισμός αυτός μας επιτρέπει ακριβώς να ενισχύσουμε τους ελέγχους για την πραγματική άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, ε, για την ενημέρωση δηλαδή των εργαζομένων μεταναστών. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του γεγονός τόσο ότι θέλουμε να έχουμε ε, ένα μηχανισμό για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να μπορούμε ε, τα όσα έχουμε σε εθνικό επίπεδο να τα μοιραζόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΝ που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο για την ίση μεταχείριση αυτών των εργαζομένων άκουσα και κάποιες ανησυχίες για την ποιότητα των θέσεων εργασίας που μπορεί να προσφέρονται μέσω του Euros. Εδώ πραγματικά θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διατίθεται αυτό το οποίο διατίθεται σε εθνικό επίπεδο. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται σε εθνικό επίπεδο, ε, μόνο που οι θέσεις εργασίας που αυτή τη στιγμή ε, εν μέρη ε, είναι γνωστές σε μικρότερο επίπεδο, θα γίνονται γνωστές σε μεγαλύτερο επίπεδο. Ο έλεγχος ποιότητας λοιπόν γίνεται μεν, αλλά γίνεται με βάση τις προδιαγραφές σε εθνικό επίπεδο, που ε, είναι ε, ήδη αρκετά αυστηρές. Η κοινωνική εταίροι, ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν, ο οποίος είναι σημαντικός, ε, συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του Γιούρες, συμμετέχουν ενεργά και είναι ιδιαίτερα δραστήριοι. Έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την προώθηση πρωτοφουλειών σε επίπεδο διαμεθοριακών περιοχών. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων διαμεθοριακών στην Ευρώπη, αρκετά εκατομμύρια και πρόκειται για μια ιδιαιτερότητα την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, το θέμα αυτό εξετάζεται και στον προπολογισμό, τον οποίο συζητήσατε πέρσι, ώστε να χρηματοδοτούνται κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένε και είναι και συμπληρωματικές ε, στα όσα κάνει το Euros. Έχουμε λοιπόν μία προσφορά, μία υπηρεσία, συγγνώμη, η οποία βασίζεται σε ένα δίκτυο ε, εταίρων και δημοσίων και ιδιωτικών που ε, δίνουν κάποια στοιχεία ελέγχου ποιότητας και κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες είναι πιο συγκεκριμένες και μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και ε, να έχουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες υπηρεσίες για τις περιφέρειες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι και σε σύμπραξη με τις εθνικές ε, υπηρεσίες και τους οργανισμούς απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Θέλουμε λοιπόν αυτή η διαμεθοριακή εταιρική σχέση να συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά τη διαφορά του σχεδίου κανονισμού και της οδηγίας για την παροχή των υπηρεσιών, η οδηγία για την άσκηση των δικαιωμάτων είναι σαφώς η οδηγία για τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων. Επομένως, την εφαρμογή των διατάξεων του 492 ε, για να μην υπάρχει ε, διάκριση για τους μετανάστες εργοζομένων και το EURES είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει να ενημερωθεί κάποιος για την προσφορά θέσεων εργασίας, για τις συνθήκες εργασίας, για τις συνθήκες οι οποίες αφορούν την απασχόληση ε, σε θέματα κινητικότητας. Επομένως, τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται. Αλλά τίποτα δεν απαγορεύει σε ένα κράτος μέλος να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις δομές οι οποίες δημιουργούνται στα πλαίσια της οδηγίας ή να εντάξει τα όσα προβλέπονται από την οδηγία ε, σε ένα δίκτυο γιούρες. Πρόκειται λοιπόν για συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία προσφέρονται σε εθνικό επίπεδο και μπορεί κάλλιστα κάποιο να τα υλοποιήσει. Όσον αφορά του στόχου όμω, οι στόχοι είναι συμπληρωματικοί επίση. Όσον αφορά την τελευταία σα ερώτηση, που αφορά το άρθρο 38 του 492, ε, να σα πω ότι το σχέδιο κανονισμού υποκαθιστά και το κεφάλαιο 2 του κανονισμού 492 ε, και το άρθρο 38 του κανονισμού και στο άρθρο 33 περιλαμβάνει πλέον διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα της ε, αρμοδιότητας εκτέλεσης και εκχώρησης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό διασκεδάζει τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ε, απόφασης του 2012. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν εδώ την ανταλλαγή απόψεων. Βλέπουμε πόσες δυσκολίες ε, θα προκύψουν και κάποιες οποίες έχουμε ήδη διαπιστώσει όταν εξετάσαμε ε, κάποιες ε, προτάσεις. Η Edith Bauer ανέφερε μία, η Γιούτα μια άλλη. Θα μπορούσα να αναφερθώ και εγώ στην πρόταση την οποία συζητήσαμε στα πλαίσια των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Υπάρχει νομοθεσία η οποία θα έπρεπε κανονικά να παρουσιαστεί ως δέσμη μέτρων και ε, λόγω επίγουσας ανάγκης ε, όλα αυτά παρουσιάζονται εμβαλωματικά και θεωρώ ότι όταν γίνει μια συνολική πρόταση μαζί με το σχέδιο κανονισμού, η διάρθρωση της συζήτησης που έγινε στα πλαίσια του προπολογισμού και των ε, πιο επιχειρησιακών στοιχείων θα μας δημιουργήσει αρκετές απορίες και κάποια προβλήματα γιατί θα υπάρχουν παρεμβάσεις μεταξύ των δύο και θεωρώ ότι θα πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο ναι, μεν πρέπει να εφαρμοστεί κατεπηγόντω, διότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και δύσκολη η διαπραγμάτευσή του, διότι βρισκόμαστε σε ένα περίπλοκο πλαίσιο από πλευρά ε, τη επίσημη παρουσίασή του και περιλαμβάνει και κάποιες σημαντικές προτάσει. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακούσαμε λοιπόν τα όλα όσα αφορούν το κείμενο αυτό. Από ό,τι κατάλαβα στο Συμβούλιο η συζήτηση προχωρά δυναμικά, για να το θέσω έτσι. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε όχι μόνο με την ημερήσια διάταξη, αλλά και τις εργασίες της Επιτροπής Απασχόλησης στη διάρκεια αυτής της 7ης θητείας. Σας καλώ λοιπόν να μείνετε στην αίθουσα για την φωτογραφία και στη συνέχεια θα πάμε έξω για το ποτό αυτό το αποχαιρετιστήριο. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ και τους διερμηνούς η Πρόεδρος που ήταν εδώ μέχρι το τελευταίο λεπτό.